Λοιπόν, liebe Kolleginnen und Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, να έρχεται και ο Σούστερ, θα ξεκινήσουμε. Χαίρομαι που τώρα, κατά την έναξη της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου, Βρίσκεται μαζί μας ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που είναι και αρμόδιος για το διεθνές εμπόριο, ο κύριος Ζων Άσελπον. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Οι προτεραιότητες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας συνδέονται με πολύ συναρπαστικά θέματα, όχι μόνο όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, αλλά και όσον αφορά την καλύτερη νομοθεσία, την ανάπτυξη, την, την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το θέμα της γειτονίας και της Ουκρανίας. όπως και η περαιτέρω εξέλιξη ε, στα πολυμερή θέματα όπως είναι οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ. Έχουμε και τρία νομοθετήματα που μας ενδιαφέρουν, τα ε, ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές ε, που από πολιτικής πλευράς είναι αρκετά σημαντικό θέμα, το θέμα της αμοιβαιότητας και προσωπικά για μένα προτεραιότητα αποτελεί το Trade Defense Instrument, ένα μέσο ώστε να μπορούμε να αντιδρούμε στη διεθνή αγορά. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι χθες ε, είχαμε μία κρόαση για ε, την διαφάνεια σε μηχανισμούς διατησίας. Στην Ουνσιτράλ, όπου προβλέπεται η διαφάνεια όχι μόνο για την νέα στη συμφωνία, αλλά και για παλαιότερες. Μέχρι τώρα, στο Συμβούλιο φαίνεται ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ε, πετύχαμε συμφωνία. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια. Αυτή ήταν η δική μου εισαγωγή. Ο κύριος Άσελπον θα μας ε, κάνει μια εισαγωγή και κατόπιν θα έχουμε τρία τέταρτα να συζητήσουμε μαζί του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε εδώ σήμερα το απόγευμα. Έχω προετοιμάσει μια εισαγωγική παρέμβαση, αλλά επειδή είμαστε όλοι πολιτικοί και επειδή είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, μετά από 13 χρόνια διαπραγμάτευσης φτάσαμε σε μια συμφωνία με το Ιράν σήμερα το πρωί στη Βιέννη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν ήδη επιπτώσεις στη τιμή του πετρελαίου. Ένα Ιράν επικοδομητικό που επανέρχεται στη διεθνή κοινότητα και που δεν είναι πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό. Οι εντάσεις ε, στον αραβικό κόσμο σήμερα οφείλονται στις διαφορές Σιητών και Σουνιτών. Και ελπίζω ότι το Ιράν σήμερα, αλλά και η Σαουδική Αραβία κυρίως, θα μπορέσουν να συμφωνήσουν για να επιλύσουν και να ξεπεραστεί αυτή η αστάθεια που υπάρχει όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά εν γέννη στο μουσουλμανικό κόσμο. Είναι η 12η Προεδρία του Λουξεμβούργου αυτή. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ, γιατί βλέπω ότι 13 κοινοβουλευτικές επιτροπές ενδιαφέρονται για κάποια προβλήματα που αφορούν συγκρούσεις κτλ. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνομιλήσω με τις επιτροπές αυτές. Δώστε μου ένα τεταρτάκι όμως πρώτα για να σας πω επίσημα τι σκοπεύουμε να κάνουμε ε, ως Προεδρία και που αφορά την Επιτροπή σας βέβαια. Στο πρόγραμμά μας έχουμε βάλει τον τίτλο Ένωση για τους πολίτες, πιο κοντά στους ε, πολίτες, στις προσδοκίες τους, τις ε, οργανώσεις τους ε, και υποστήριξη των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δική μας Προεδρία, με βάση την παράδοσή της που έχει και τις πεπιθήσεις της, θα προσπαθήσει να βάλει τους πολίτες στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Πολύ περισσότερο σήμερα παρά ποτέ θέλουμε τα πραγματικά και άμεσα συμφέροντα των πολιτών να λαμβάνονται υπόψη σε όλε τι ενωσιακέ πολιτικέ. Γι' αυτό βασιζόμαστε σε εσά για να υπερασπιστούμε μια εμπορική πολιτική ευρωπαϊκή που συμπεριλαμβάνει όλου, ε, λογική, συνεπή, που δίνει πραγματικέ ευκαιρίε ε, πρόσβαση στι αγορέ των χωρών εταίρων. Αν το Λουξεμβούργο θέλει να δημιουργήσει ανοιχτά εμπορικά ε, περιβάλλοντα, δίκαια, που προωθούν τι θέσει απασχόληση, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Από την άλλη όμω ξέρουμε πολύ καλά τι απαιτήσει και τι προσδοκίε έχουν οι εταίροι μα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων, κάποια ευαίσθητα θέματα επίση που του απασχολούν που αφορούν τι επενδύσει ή την διασφάλιση των κοινωνικών ρητρών και περιβαλλοντικών ρητρών. Και εμεί κυρίω θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε σε τρίτε χώρε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να έχουμε έναν μόνιμο διάλογο μεταξύ ε, του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν, του Συμβουλίου και της Κοινωνίας των Πολιτών. Ε, αυτές οι πολιτικές σε διάφορα επίπεδα αυτό ακριβώς προωθούν. Ε, και ε, το εμπόριο, ε, βιομηχανία, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες πολιτικές. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, Πρόεδρε, με αυτό το πνεύμα να καθοδηγήσουμε τις πολιτικές μας τους επόμενους 6 Θέλουμε να ενταχθούμε σε μια έτσι ρεαλιστική παράδοση, πραγματιστική, ε, να υπάρξει συνέχεια και να ακολουθούν το καλό παράδειγμα των ε, συναδέλφων των Λετώνων που τους χαιρετίζω εδώ γιατί έκαναν μια θαυμάσια δουλειά το πρώτο εξάμεινο του 2015. Πριν μπω σε συγκεκριμένα ντοσχέ και μιλήσω για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις αλλά και διμερείς αλλά και για τα νομοθετικά κείμενα που προωθούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα σημαντικό ε, για τη σημασία που έχει μια καλή εμπορική πολιτική που συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Μην ξεχνάτε την ε, δολοφονική επίθεση που έγινε στην Τινησία, που αφορούσε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα. Η χώρα αυτή εξαρτάται από τον τουρισμό, γιατί 12% του πληθυσμού, του ενεργού πληθυσμού, δουλεύει στον τουρισμό. Είναι σαφές ότι η οικονομία της Τινησίας βρίσκεται αποσταθεροποιημένη πάλι και έχει επιγόντως ανάγκη να διαφοροποιηθεί, να κινηθεί προς άλλους τομεί ε, και να αναζητήσει και άλλες γεωγραφικές αγορές. Η εμπορική πολιτική της Ένωσης μπορεί να τη βοηθήσει εδώ για να βελτιώσει τις προοπτικές θέσεων απασχόλησης, κυρίως των νέων της Τινησίας. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που επί προεδρίας μας θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία πλήρη, ενδελεχή ε, με τη χώρα αυτή, με την Τινησία. Στην, ε, στο Μαρόκο τώρα Θέλουμε να υποστηρίξουμε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και να τους δώσουμε προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ε, στα πλαίσια μιας ε, πολιτικής γειτονίας συνεπούς ε, και σε οικονομικό επίπεδο και σε εμπορικό επίπεδο. Δεν υπάρχει λόγο να σας πω ότι το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε αυτές τις χώρες να τις σταθεροποιήσουμε σε μια περιοχή όπου είναι πολύ αποσταθεροποιημένη και να του εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση θα σα μιλήσω για την ε, μελλοντική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εμπόριο που θα ανακοινωθεί, που θα εκδοθεί, αν δεν απατώμε, το φθινόπρο που μας έρχεται. Ίσως δεν είναι το πιο αγαπητό θέμα των ΜΜΕ, αλλά αυτή η στρατηγική θα, καθορίσει την πορεία της εμπορικής μας πολιτικής στα επόμενα πέντε χρόνια. Και Θέλω να πω δύο λόγια. Η τελευταία ανακοίνωση της Κομισιόν ήταν το 2010. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γενικής ε, Διεύθυνσης Εμπορίου τότε ήταν να κάνουν διαπραγματεύσεις φιλόδοξες σε όλα τα επίπεδα, ε, διμερές, πολυμερές κτλ. στη γειτονία μας αλλά και πέραν αυτής. Ε, παρατηρήθηκε ή μάλλον μετά ακολουθήθηκε από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας και την εφαρμόσαμε στη θήκη τη Λισαβόνα και στην εμπορική πολιτική. Μα επέτρεψε λοιπόν να εμβαθύνουμε τι στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να ισχύσουμε τι οικονομικέ διμερεί σχέσει τη Υπήρου μα, να υπερασπιστούμε τι αξίε μα και τα συμφέροντά μα. Ξεκινήσαμε να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα βιώσιμη ανάπτυξη, ε, στην πρόσβαση των εμπόρων μα και των μικρομεσαίων μα επιχειρήσεων σε τρίτε αγορέ και στο σεβασμό την, τον κανόνα πνευματική ιδιοκτησία. Πολλά θέματα προωθήθηκαν και εσωτερικά για να μεταρρυθμίσουμε, παραδείγματο χάρη, την αμυντική εμπορική μα πολιτική. Παρά τα όσα έχουμε κάνει, παραμένουν πάρα πολλά που δεν έχουμε κάνει και η νέα ε, εμπορική στρατηγική που θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο θα προσανατολιστεί σίγουρα σε αυτού του στόχου. Ορισμένοι δεν έχουν υλοποιηθεί εξάλλου, ενώ κάποιε άλλε προκλήσει έχουν εμφανιστεί στο μεταξύ το 2010 και σήμερα, μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ κρατών μελών πιο ευρέω την ε, θεώρησή μα για την νέα εμπορική πολιτική προσαρμοσμένη στι ανάγκε. Ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων Εμπορίου θα υιοθετήσει συμπεράσματα ε, στην συνεδρίαση τη 27η Νοεμβρίου. Ε, πολυμερή θέματα. Η ΟΠΟΕ θα συνεδριάσει, όπως ξέρετε, στο Ναϊρόμπι το Δεκέμβριο. Η δέκατη Υπουργική Σύνοδο θα είναι αυτή. Και η ατζέντα αυτή, η διμερής, είναι πάρα πολύ βεβαρημένη. Θα επανέλθω σε μια στιγμή. Αλλά και το πολυμερές πλαίσιο παραμένει για τη χώρα μας βασικό στοιχείο και για την εμπορική πολιτική. Χωρίς σαφείς κανόνες ε, σε πολυμερές επίπεδο η παγκοσμιοποίηση θα γινόταν ένα χάος και πολύ πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι, ανα... και οι χώρες και οι αναπτυγμένες χώρες οι χώρες του Βορρά, οι χώρες του Νότου αδύνατο να συμφωνήσουμε το εμπόριο δεν είναι μία καθαρόεμη τέχνη. Δεν γίνεται, δεν αφορά μόνο κάποιες βιομηχανικέ, εκβιομηχανισμένε ας πούμε και προηγμένε χώρε. Είναι εργαλείο το εμπόριο. Για όλου. Και για τους πολίτες, καθώς και αυτού που ζουν πέρα από τα σύνορά μα, που θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο αυτού του πλανήτη και να πετύχουμε μια ανάπτυξη πολυμερή. Το 2001 στον κύκλο της Ντόχα, όταν ξεκίνησε ο κύκλος της Ντόχα, θέλαμε να εντάξουμε περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες σε μια οικονομία σε μόνιμη αλλαγή μέσω εργαλείων ευελιξίας για τους πιο ενδεείς, μείωση των ε, τελωνιακών δασμών, που μπλοκάρει τις εξαγωγές ειδικά των ε, αναπτυσσόμενων χωρών. Ε, σήμερα τα περισσότερα μέλη του ΠΟΕ είναι αναπτυσσόμενες χώρες και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο αριθμός των προσχωρήσεων των ε, λιγότερων επιτυχμένων χωρών στον ΠΟΕ είναι πραγματικά μια success story. Το συμπέρασμα και μετά από δύο χρόνια που συμφωνήθηκε η Συμφωνία διευκόλυσης των Συναλλαγών και η τομεακές εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ο μιλητής ε, διορθώνει ότι άλλαξαν οι νοοτροπίες στις λιγότερες, ε, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χάρη στον ΠΟΕ και χάρη στις διαπραγματεύσεις που γίνονται επίσης. Αλλά αυτή είναι η αρχή. Μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να προετοιμάσουμε το έταφος ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο κύκλος της Ντόχα το να συνεχίζονται ατέρμονα αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι κατά της αξιοπιστίας του ΠΟΕ και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χάνουν ευκαιρίες για να συμμετάσχουν καλύτερα στις ε, παγκόσμιες ροές, στις παγκόσμιες συναλλαγές και στις παγκόσμιες επενδύσεις. Ποιο λόγια για τη συμφωνία για την διευκόλυνση των συναλλαγών. Το Συμβούλιο ε, βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε η επικύρωση Τη λεγόμενη της λεγόμενης συμφωνίας να γίνει μέχρι τον Οκτώβριο αν γίνεται. Και έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταθέσει το εργαλείο προσχώρησης στη συμφωνία πριν από την Υπουργική του Ναϊρόμπι. Στα περιθώρια της 10ης ε, Υπουργικής Συνόδου στο Ναϊρόμπι ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε σε πολιτικό επίπεδο τη συμφωνία πολυμερούς χαρακτήρα για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Αυτή η συμφωνία εντάσσεται και αυτή σε μια λογική μεγαλύτερη έτσι, συνέπεια τη εμπορική μα πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, βιομηχανική πολιτική και καινοτομία. Οι διαπραγματευτέ ασχολούνται αυτή τη στιγμή σε ένα πρωτόλιο τη συμφωνία και οι συζητήσει θα γίνουν και για το οριζόντιο κείμενο τη συμφωνία που θα αφορά και το θέμα των υπηρεσιών και των μη δεσμολογικών φραγμών. Αυτή η συμφωνία θα είναι πολύ σημαντική και στο πλαίσιο των κλιματικών διαπραγματεύσεων COP21 στο Παρίσι και της υπουργική του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι. Η συμφωνία θα είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα και θα είναι επωφελές αυτό για την Ευρώπη και για τους ε, εταίρους σε διάφορα επίπεδα, το περιβαλλοντικό, ε, κοινωνικό, οικονομικό κτλ. Πέρα από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις υπάρχει ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή για την αναθεώρηση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ελπίζουμε όμως να υπάρξει θετική εξέλιξη τις ε, επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία ΤΙΖΑ, η Λουξεμβουργία και η Προεδρία θα παρακολουθήσει το πώς εξελίσσεται το πράγμα στο, στο εσωτερικό του Συμβουλίου και αν η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω ε, ενός διαφανούς ε, εμπορικού εργαλείου μη διακριτικής μεταχείρισης, αν γίνουν όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την... Ε, θα, προ... είναι πολύ θετικό αυτό για αυτούς τους τομείς. Η υπηρεσίε θα αποκλειστούν από τι διαπραγματεύσει και το θέμα της προστασία της ιδιωτική σφαίρας θα διατηρηθεί. Επίσης, στο Συμβούλιο θα υποστηρίξουμε τι ε, διαπραγματεύσει και θα συνεργαστούμε στενά με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε η εκφώνηση νέων κανόνων ε, για τι υπηρεσίε με σεβασμό των, ε, του κοινοτικού κεκτημένου να δώσουν νέες ευκαιρίες στους προμηθευτές υπηρεσιών στους παρόχου υπηρεσιών. Τώρα θα ήθελα να μπω στι διαπραγματεύσεις για τις διμερείς, να μπω ε, διαπραγματεύσεις. Θα προσπαθήσουμε η διαπραγματεύση για τη Συμφωνία ε, Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης, ε, το TTIP δηλαδή, για το εμπόριο και τι επενδύσει, να φτάσει σε ένα νέο επίπεδο ε, σε ό,τι αφορά την ουσία, το διάλογο και τη διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο δεύτερο γύρος διαπραγματεύσεων ε, στις Βρυξέλλες και Ξέρουμε ότι οι επόμενες εβδομάδε και μήνες θα είναι αποφασιστικοί για να καθορίσουμε την οδό που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον για τα πιο πολιτικά θέματα, τα κανονιστικά θέματα, τις υπηρεσίες, την βιώσιμη ανάπτυξη ε, και τις ε, δημόσιες προμήθειες στην Αμερική. Η Προεδρία θέλει ε, να βοηθήσει για να υπάρξει μια μεταρρύθμιση του κανονισμού ISDS που είναι η ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Το Κοινοβούλιο παίζει θετικό ρόλο στι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και κυρίω την Επιτροπή σα, την Επιτροπή ΙΝΤΑ, για το ψήφισμά σα που θα μα επιτρέπει να ενισχύσουμε τη θέση τη διαπραγματεύση με τι ΗΠΑ και να προχωρήσουμε στη συζήτησή μα. Το Λουξεμβούργο θα είναι στη διάθεσή σα, ούτω ώστε να συζητήσουμε αυτό το πολύ αμφίσιμο, ε, και επίμαχο σημείο. Υπάρχουν κάποιες κριτικές για αυτέ τι διαπραγματεύσει, Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτές. καταλαβαίνω αυτέ τι επικρίσεις και καταλαβαίνω ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά την ε, υπόθεση του NSA σε καμία περίπτωση δεν άφησε την ε, εμπιστοσύνη της ε, κοινωνίας των πολιτών στη σημασία των σχέσεων με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κι όμω είμαι πεπισμένο ότι επειδή ο κόσμο είναι πολυπολικό και και επειδή έχουμε στενέ σχέσει με την Αμερική, μια τέτοια πλήρη συμφωνία και ποιοτική συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα τη λύση και να μα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση μεν των δε. Το είπα και το είπα πολλέ φορέ. Το κοινοβούλιο μα, στο κοινοβούλιο μα ε, στο Λουξεμβούργο, εμεί δεν θέλουμε ένα τύπ δε και καλά. Μία ε, συμφωνία με τι αξίε όμω τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν κάτι τελείω διαφορετικό από μία συμφωνία χωρί την Ευρώπη. Ένα TTIP χωρί την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το ανοιχτό πνεύμα συνεχίζουμε τη συζήτηση με όλου του εμπλεκόμενου φορεί και το Λουξεμβούργο θα οργανώσει μια διάσκεψη για το θέμα του TTIP στι Βρυξέλλε με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Εμπόριο Νοέμβριο 2015 στη Βορειοαμερικανική Ήπερο έχουμε ολοκληρωθεί από δύο χρόνια μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά, τη συμφωνία ΣΕΤΑ και έχει βγει αυτή η συμφωνία. Το νομικό χτένισμα είναι στην τελική ευθεία και θα αποφασίσουμε την κατάλληλη στιγμή πότε θα υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία που το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι ε, επιμερισμένη αρμοδιότητα στα εθνικά μα κοινοβούλια. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφαθούν για τη συμφωνία αυτή όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η Προεδρία έχει λάβει ε, πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες. Μια άλλη Προεδρία της ε, Προεδρίας μας, σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμφωνίες, ε, είναι ότι θα ε, εντατικοποιήσουμε τις ε, συνομιλίες μας για να έχουμε μια ε, φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ε, Ιαπωνία. Αυτό το ξαναείπαμε στην Σύνοδο Κορυφής 29 Μαΐου, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. αυτό το Λουξεμβούργο θα θα πλαισιώνει επικοδομητικά τις συζητήσεις για τις δημόσιες προμήθειες, για τις μη δασμολογικές ε, τροχοπέδες, μη φραγμούς ε, και τα, την πνευματική διοκτησία. Παράλληλες διαπραγματεύσεις γίνονται ε, για το TTP, που είναι η, η ειρηνική συμφωνία με τις χώρες του ειρηνικού, δηλαδή η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα εξασφαλίσει την καλή εξέλιξη των τελευταίων φάσεων των διαπραγματεύσεων με, την, ε, με το Βιετνάμ για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη χώρα αυτή. Ε, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή πολύ σύντομα. Ε, πρέπει να επιληθούν τα τελευταία ανοιχτά θέματα με την αδειόμενη αυτή χώρα στην Ασία και μάλιστα στην Νότια Ανατολική Ασία. Η συμφωνία αυτή θα είναι τέλειο προηγούμενο για άλλους τρίτους εταίρους, για άλλες χώρες στην περιοχή για την απελευθέρωση των δασμών, ε, σεβασμό της πνευματικής μας ιδιοκτησίας ε, και σεβασμό των διατάξεων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Χαίρομαι που το Βιετνάμ από επί χρόνια ήταν μία από τις χώρες όπου εμείς ως Λουξεμβούργο δίναμε αναπτυξιακή βοήθεια. Ετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε τη χώρα αυτή ε, διμερή συμφωνία ως Ευρωπαϊκή Ένωση πια όμως. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε που εμβαθύνουμε και τι οικονομικέ μα σχέσει ε, με την ΑΖΕΑΝ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΖΕΑΝ, αλλά και Ευρωπαϊκή Ένωση με την κάθε μία από τι χώρε αυτέ. Ε, με τη Μαλαισία ειδικά. Ε, και περιμένουμε την πολιτική μετάβαση με την Ταϊλάν δηλαδή για να ξαναρχίσουμε τι διαπραγματεύσει με τη σημαντική αυτή χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης, παρακολουθούμε εκ του ε, τις διαπραγματεύσεις ε, για, για τις επενδύσεις με τη Μιανμάρ και την ε, Κίνα, ούτως ώστε να προσφέρουμε βελτιωμένη προστασία των ε, Ευρωπαίων επενδυτών στις χώρες αυτές. Θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου και θα μειωθούν τα εμπόδια για τις επενδύσεις. Η δίκαιη μεταχείριση των επενδυτών και η αύξηση των επενδυτικών ροών και προ τι δύο κατευθύνσει είναι βασικό στοιχείο των δύο συμφωνιών αυτών και η Ξεβουλία και η Προεδρία θα διεκδικεί μία φιλόδοξη προσέγγιση ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, και άλλοι ασιάδε εταίροι πρέπει να αναφερθούν η Νέα Ζηλανδία και η Ζηλανδία Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία λοιπόν θέλουμε να κάνουμε όχι μόνο εμπορικέ ε, διαπραγματεύσει. Του επόμενου μήνε. θα δούμε τι απαραίτητε παραμέτρου για να δούμε τι είδου διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουμε. Επίσης, περιμένουμε να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις ενδεχομένως ε, με μια πολύ σημαντική χώρα, την Ινδία. Το μπλοκάρισμα των διαπραγματεύσεων ε, πριν από τις τελευταίες ειδικέ εκλογές δεν έχει επιληθεί ακόμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με το νέο Δελχή. Μεταξύ των ε, υπαρχουσών ε, συμφωνιών θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία με το Μεξικό και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορέσουν να γίνουν για αυτό το λόγο το συντομότερο δυνατόν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθούμε τη διαδικασία scooping που γίνεται με τη χιλή, ούτω ώστε να βελτιώσουμε αμοιβαία τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που χρονολογείται το 2002. Στη Λατινική Αμερική επίσης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να οριστικοποιήσουμε την προσχώρηση του Εκουαδόρ στην ζώνη ελευθέρων συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολομβίας, Περού. Και θα αναφερθώ και στο Μερκοσούρ, Βραζιλία, Αργεντινή δηλαδή, Παραγουάι Ουρουγουάη και Βενεζουέλα, όπου παρά τις προσπάθειές μας οι διαπραγματεύσεις ε, πόρα απέχουν από το τελικό του σημείο και περιμένουμε την προσφορά του Μερκοσούρ μέχρι το τέλος 2015. Άλλες προκλήσεις μας ε, περιμένουν ε, στην ε, ανατολική μας γειτονία, κυρίως η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ε, με την Ουκρανία, που θα τεθεί σε ισχύ 1η Ιανουαρίου του 2016, σε αυτό το πλαίσιο οι Ευρωπαίοι ε, εμπειρογνώμονε, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονε θα συνεχίσουν τι συζητήσει σε επιμερέ επίπεδο για να αποφύγουμε αυτή η συμφωνία να οδηγήσει σε μια επιδείνωση περαιτέρω τη πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία. Ο διάλογο θα πρέπει να συνεχίσει με σεβασμό των συμφερόντων διαφόρων μερών και των κυρίαρχων επιλογών των ε, εταίρων. Αυτές οι διαβουλεύσεις δεν αρέσουν σε όλους, το ξέρω, αλλά θα πρέπει να παραμένουμε και ανοιχτοί στην προσέγγιση μας και να τίνουμε ευηκοούς τις απόψεις τους. Η Ρωσία, χωρίς ε, καμία αμφιβολία, θα ενισχύσει έτσι τις ε, οικονομικές σχέσεις στην Ήπειρό μας και μέσω εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Την Μολδαβία και τη Γεωργία. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να εμβαθύνει αυτέ τι οικονομικέ σχέσει ανά περίπτωση με τι χώρε γειτονία. Υπενθυμίζω ότι η Κομισιόν ε, έκανε μια πρόταση κανονισμού σε ό,τι αφορά την ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μηχανισμού κατά της, ε, του λαθρεμπορίου στην συμφωνία με τη Μολδαβία καθώς και στη Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωση Γεωργίας. Η Προεδρία μας θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ε, νομοθετική διαδικασία σχετικά με αυτό το θέμα ε, και θέλουμε να φτάσουμε και σε θέση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Θα, θα ακούσουμε την άποψη του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά και πιστεύουμε ότι θα ξαναρχίσουν γρήγορα οι τριμερείς διάλογοι. Θα πρέπει να πάρουμε σύντομα αποφάσεις για να εγκρίνουμε την ε, προσχώρηση του Καζακστάν στο ΠΟΕ και συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη χώρα αυτή. Η Προεδρία μας θα θελήσει να δώσει το Συμβούλιο διαπραγματευτική εντολή για μια συμφωνία α, μη προτιμησιακής μεταχείρισης με την Αρμενία. Θα προωθήσουμε τους προτιμησιακούς εμπορικού δεσμούς με τους Αφρικανούς εταίρους. Για μας οι οικονομικές ε, ε, συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης είναι ευκαιρία για τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές και μπορούμε να τις βάλουμε και σε μια νέα βάση ε, θα πρέπει να έχουμε μια συνεπή πολιτική στην Αφρική, όπου βέβαια αντιμετωπίζουν ε, πάρα πολλέ προκλήσει, αλλά υπάρχουν και πολλέ ευκαιρίε. Το εμπόριο εδώ θα πρέπει όχι μόνο να εξυπηρετεί την ανάπτυξη οικονομική πίσω των μετέρων μα, αλλά θα πρέπει να μα βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα εμένα του δε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την κοινωνία. Στα πλαίσια μια στενή εταιρική σχέση μεταξύ των δύο υπήρων. Τέλο, θα ήθελα να μιλήσω για η συνομοθετική διαδικασία. Μία από τι προτεραιότητε τη Προεδρία μα θα είναι η πρόταση κανονισμού για τα μέταλλα, μεταλλεύματα από περιοχέ κινδύνου για να αυξήσουμε την ε, ασφάλεια δικαίου και την ε, διαφάνεια στην αληθινή εφοδιασμού για να σπάσουμε δεσμό ανάμεσα στην εξόριξη των μεταλλευμάτων, το εμπόριό του και τη χρηματοδότηση των ε, πολέμων και σειράξεων. Το Η Κοινοβούλη ψήφισε τροπολογίε σε αυτή την πρόταση στη σύνοδο του, 20ης Μαΐου η Προεδρία μας θα προσπαθήσει να κάνει καλές και προβληματικές συζητήσεις στο Συμβούλιο, ώστε να ολοκληρώσουμε την πρόταση των 28 χωρών. Λαμβάνοντα υπόψη τι τροπολογίε που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο στόχο μα θα είναι να βάλουμε να πετύχουν μια πραγματευτική εντολή του Συμβουλίου, τόσο ώστε να ξεκινήσουμε το τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, θα πρέπει αυτό ο κανονισμός να τεθεί σε ισχύ ούτω ώστε να υποφεληθούν οι πληθυσμοί και οι τοπικέ κοινότητε και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στι πρώτε ύλες ε, Εμεί, ε, οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι δηλαδή οι προμηθευτέ, με διαφάνεια και σεβασμό του διεθνούς, των διεθνών κανόνων. Το να φύγει κάποιο από μια περιοχή και να μπει κάποιο άλλο στη θέση του δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είναι καλό ούτε για τι χώρε ούτε για του εμπορευομένου μα. Μια συνεπή πολιτική είναι το κλειδί και αυτό θα προσανατολίσει τη στάση στην Προεδρία μας. Επίσης, η τροπολογία του κανονισμού για το εμπόριο κάποιων αγαθών το, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή ή για το βασανιστήρια. Ο κανονισμός υιοθετήθηκε από τη Λουξεμβουργία της Προεδρίας πριν από 10 χρόνια, το 2005, και μας ενδιαφέρει τα μάλα. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για τις τροπολογίες που προτάθηκαν από την Κομισιόν έχουν προχωρήσει και χαιρόμαστε εκ των προτέρων που θα ακούσουμε και την άποψη του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Η η Προεδρία έχει σαν στόχο να φτάσουμε σε μια εντολή του Συμβουλίου για την πρόταση αυτή και να μπούμε σε τριμερή διάλογο με το Κοινοβούλιο και να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης μέχρι το τέλος του 2015 αν γίνεται. Φυσικά, μετά είναι οι Ολλανδοί, έτσι. Καλή προεδρία θα είναι και αυτή. Φυσικά, Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο περιμένει την αντίδραση του Συμβουλίου στο φάκελο για τον ε, εξυγχρονισμό των αμυντικών εμπορικών εργαλείων. Το anti-dumping δηλαδή. Το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση τον Απρίλιο του 2014, αλλά τα κράτη-μέλη είναι διαιρεμένα για το θέμα των κανόνων και η συζήτηση του Ανατολισμού στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στι 20, 21 Νοεμβρίου του 2014 δεν μας επέτρεψε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Η Προεδρία μας είχε μία ενδιάμεση θέση στις συζητήσεις στο Συμβούλιο και είναι έτοιμη βεβαίως να διερευνήσει διαφορετικές συναλλακτικές λύσεις για να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Και επίσης περιμένουμε μια ανάλυση της Κομισιόν ε, για το θέμα της Κίνας και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε στη σχέση μας με την Κίνα. Αυτά θα δουλέψουμε εργοδός. Δεν πρόκειται να σταυρώσουμε τα χέρια όπως βλέπετε. Θα είμαστε στην ε, διάθεσή σας, θα σας ακούσουμε και χαιρόμαστε που μπορούμε να δουλέψουμε καλά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Merci euh, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Για την συζήτηση προτείνω πεν, δύο λεπτά ο κάθε ευρωβουλευτής τη παρεμβάση. Η κυρία Ρέντινγκ είναι η πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λεπτά αδύνατον. Ακόμα και αν είμαι ταχύτατη, δεν μπορώ να ολοκληρώσω δύο λεπτά. Εν ονόματι του ΕΛΚ, θέλω να σα ευχαριστήσω, Πρόεδρε, για όλε τι λεπτομέρειε που μα δώσατε για τα σημερινά και μελλοντικά project. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη ενοποίηση. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και στο εξωτερικό εμπόριο πρέπει να δημιουργήσουμε διεθνείς κανόνες καλούς και να εφαρμόσουμε να δημιουργήσουμε προσκόμματα σε αυτή την κούρσα προς τα κάτω που γίνεται. Εάν διαβάσω τα προγράμματα της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, τι βλέπουμε ως λέξη κλειδιά. Συνέχεια και συνέπεια. Χρειάζονται αυτά, αλλά δεν αρκούν. Επιτρέψτε μου να δούμε καταρχάς τη συνέχεια. Το θέμα της συνέχειας. Τι είπατε, Πρόεδρε, ότι η Κομισιόν εκπονεί την νέα της έκθεση για το μέλλον του εξωτερικού εμπορίου. Για να υπάρχει συνέχεια, θα πρέπει συνέχεια να διαπραγματευόμαστε με τους συνήθεις υπόπτους ε, για τα συνήθεις θέματα. Έχει νόημα αυτό. Ή μήπω πρέπει να συζητήσουμε με νέους εταίρους για νέα θέματα. Παραδείγματο χάρη με τους BRICS και τους MINT. Γιατί εκεί υπάρχουν οι εμπορικοί ε, φραγμοί. Και εκεί όμως υπάρχει και το δυναμικό ανάπτυξη το πιο υψηλό. Μήπως λοιπόν η η Προεδρία θα έπρεπε να αλλάξει προτεραιότητε τη σε αυτό το θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ό,τι αφορά το ΤΙΖΑ είπατε και κάτι προφορικά τώρα. Γιατί στο πρόγραμμά σας το θέμα αυτό δεν αναφέρεται καθόλου. Όμως, Υπάρχουν πολλέ χώρε που διαπραγματεύονται μαζί μα, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένε Πολιτείε, και που θεωρούν ότι είναι προτεραιότητά του. Επίση, το θέμα του, της, των πολυμερών διαπραγματεύσεων είναι μεγάλη πρόκληση. Και θα είναι και μάλιστα και ένα εφαλτήριο, αν θέλετε, για να δούμε αν θα πρέπει να πολυμερίσουμε εντό αγωγικών τις προσπάθειές μας στο μέλλον. Ίσως αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε ενώπιση του Ναϊρόμπι. Μιλήσατε επίσης για συνέπεια. Χρειάζεται συνέπεια, προφανώς. Γιατί? Γιατί τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται οι διαπραγματεύσεις, τι συνέπεια υπάρχει σε διεθνές επίπεδο. Ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη μία έχουμε το Συμβούλιο και από την άλλη έχουμε το Κοινοβούλιο και υπάρχει γενική κακοφωνία και σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των πολιτών, των τοπικών αρχών κτλ. Απόλυτη κακοφωνία. Θέλουμε να πάρει θέση η Κομισιόν εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία εδώ. Σπάνια τίθεται αυτό το θέμα. Οι φυσικοί φραγμοί εξαφανίζονται. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται να τους αντικαταστήσει με ένα μοσαϊκό κανονιστικών κανόνων. Θέλουμε περισσότερη, δηλαδή επιβάλλουμε περισσότερη γραφειοκρατία, όλο και περισσότερη γραφειοκρατία. Εμείς θέλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγκόσμια έτσι, ισοτιμία, level playing field. Είπαμε εμείς το τι ας πούμε, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Τι πιστεύει η Προεδρία σας γενικά το Συμβούλιο θα το συζητήσει αυτό το θέμα. Επίσης, τι γίνεται με το ISDS, τι γίνεται με το Μηχανισμό Επίλυσης ε, Διαφορών Επενδυτών Κράτους. Το Κοινοβούλιο θα σαφές για αυτό το θέμα. Περιμένουμε υπό την ηγεσία σας τη θέση του Συμβουλίου για το ISDS. Και περιμένουμε τη διάσκεψη με τους κοινωνικούς εταίρους. Την περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Α, μάλιστα. Τη θέλουμε τη διαφάνεια. Όμως, γιατί εδώ έχουμε διαφάνεια στο, στο χ σημείο, ας πούμε, και όχι στο ψ σημείο. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας συνεπής. Ε, άλλα υπάρχουν για το τίσα, άλλα για το TIPA. Ε, για το τύπα έχουμε position paper για κάθε κεφάλαιο. Ενώ για το τίσα, έχουμε το Wikileaks, τίποτα άλλο. Το Wikileaks. Και για τα νομοθετικά θέματα. Γιατί το άνοιγμα των δημοσίων αγορών, ας πούμε, στις τρίτες χώρες. Η θέση της Κομισιόν είναι σαφής εδώ. και το Κοινοβούλιο. Αλλά το Συμβούλιο στηρίζει γενικθείω. Μπορεί να πιέσετε τελικά και το Συμβούλιο να πει και αυτό κάτι. Γιατί βλέπουμε σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε, χάνουμε τελικά στην αμοιβαιότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι και καινή ώρα αυτή η αρχή τη ε, ε κάπου να εγγραφεί και να την εξασφαλίσουμε βλέπω ότι ο πρόεδρος ε, σηκώνει αυτό το εργαλείο βασανισμού του. Έχω άπειρες ακόμα ερωτήσεις και το ΕΛΚ βασίζεται στην Λουξεμβουργιέζικη Προεδρία ούτως ώστε αυτά τα ερωτήματα να μπουν στο τραπέζι του Συμβουλίου επιτέλους και επιτέλους να δοθούν απαντήσεις από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε. παρακαλώ. Ο David Μάρτιν. Ερωτήσεις ε, σε σχέση με τον τόσο χρόνο από πλευράς του ΕΛΚΑ υποχρεωτικά θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε σχέση με το ψήφισμα της σύμβαση που αναφέρατε στην αρχή πρόεδρε. Είναι σημαντικό η Προεδρία να πάρει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που πίεσε να περάσει το θέμα της διαφάνειας όσον αφορά το κράτος επενδυτή στη συνέχεια δεν ήταν σε θέση να υπογράψει αυτή τη σύμβαση, σύμβαση λόγω εσωτερικών διενέξεων και διαφορών για θέματα αρμοδιοτήτων. Δεν δίνει καλή εικόνα αυτό από πλευρά μας. Όταν ζητούμε να υπάρξει κάτι, η διεθνής κοινότητα το εγκρίνει και μετά δεν υπογράφουμε λόγω εσωτερικών διενέξεων και τριβών. Είναι ικτρή κατάσταση. Πραγματικά σας ζητώ να εγγράψετε αυτό πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου για να διευθετείτε κάτι τέτοιο. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ρέντινγκ όμως ε, το, ε, ότι το Συμβούλιο δεν είναι δυνατόν να, επιστρέψει ώστε τα θέματα και τα έγγραφα να είναι ε, απόρριτα και υποεχεμήθεια όσον αφορά τις ε, συμφωνίες εμπορίου και θα πρέπει να κάνει κάτι το Συμβούλιο να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ ήταν κάπως ενηγματικό από πλευρά σας όταν είπατε ότι έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε εγκρίνουμε σε σχέση με τα προβληματικά όρικτα θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω των πολιτικών Ίσως αυτό στοχεύει στο να είναι ένα σχόλιο αυτών που εγκρίθηκαν στο Κοινοβούλιο, ίσως στοχεύει σε ένα τριμερή διάλογο, ίσως για την εντολή που αφορά αυτό το θέμα. Γιατί καταλήγουμε σε αυτή τη θέση, θα ήθελα να το γνωρίζω αυτό. Πολύ σύντομα για άλλα θέματα τώρα, για τον Καναδά. Έχετε απόλυτο δίκιο και πάλι. Αλλά όμως είσαστε και ενηγματικός κάπως όταν είπατε το κεφάλαιο για τις επενδύσεις θα μπορούσε ίσως να είναι πρόβλημα ναι, θα μπορούσε να είναι πρόβλημα, αλλά θα ήθελα να συνεχίσει να πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Προεδρία του Λουξεμβούργου όσον αφορά το θέμα ΣΥΤΑ να βελτιωθεί το κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Διότι αυτό θα διευκόλυνε το να εγκριθούν τέτοια θέματα από το Κοινοβούλιο για παράδειγμα. Ολοκληρώνω για τα προστατευτικά μέτρα για το εμπόριο. Ελήφθη το μήνυμα, είναι όμως δυσκολή, σχεδόν ανέφικτο να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο, προσπαθήστε όμως κάτι να γίνει κατά το επόμενο εξάμεινο. Πρόεδρος, πράγματι σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμπάτη παρακαλώ. Yeah, Μάλιστα, ε, Υπουργέ, ένα ευρύτατο πρόγραμμα εργασιών μας παρουσιάσατε και πολλά τέτοια κλώσματα και νήματα βρίσκονται στα χέρια σας, πώς θα τα συνθέσετε όλα αυτά πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρθηκαν θέματα τριβών στο Συμβούλιο και επιμέρους προβλήματα τα οποία αφορούν κάποιες συμφωνίες. Απλά και μόνο θα έδινα τη Συμβουλή η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κάπως πιο γενναιόδορη αν γίνεται. Για παράδειγμα χώρες όταν επιμένουν κάποια πράγματα να τα περάσουν και θέλουν να γίνει ίσως κάτι διαφορετικό, καλό είναι να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα. Γιατί το λέω αυτό. Πρώτον, είναι μια μεγάλη αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε σε σχέση με τους ε, όσους υποβάλλουν τέτοιες προσφορές οι μεγάλες, οι μεγάλες χώρες μπορούν ε, να βρουν λύσεις, οι μικρές όχι. Θα πρέπει εδώ να δούμε την πίεση που υφίσταται για μικρότερες χώρες. Και το επόμενο είναι αν θέλουμε να υπάρξει μια ανταπόκριση και να είμαστε πιο φιλελεύθεροι σε σχέση με εταίρους, αυτό δεν είναι ζημιογόνο. Αυτό κινητοποιεί την παραγωγικότητα αν πρέπει κανείς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες. Η ε, Γερμανία είχε ε, προβλήματα με τις αναβαθμίσεις, τώρα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχει η ανάγκη να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους και τους ανταγωνιστές αν υπάρχουν τριβές ή προβλήματα δεν θα πρέπει με βίαιο τρόπο να προσπαθούμε να τα επιλύσουμε αλλά θα πρέπει να γίνεται η προσπάθεια με ένα γενναιόδωρο τρόπο αντιμετώπισης να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ένα ελεύθερο πλαίσιο εμπορίου θα μπορεί να ε, υφίσταται για ε, εκείνους που μπορούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δράσουν. Ευχαριστώ. Ah, okay. Πολύ καλά. Εσείς. Η συνάδελφος θα πάρει τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Υπουργέ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας σας. Έχοντας παρακολουθήσει τα όσα αναφέρατε, θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα προκλητικές οι επόμενες εβδομάδες και μήνες. Υπάρχουν κάποια ορόσημα στην Προεδρία σας, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα τουλάχιστον. Πρώτον, η διάσκεψη του ΠΟΕ και με χαρά άκουσα ότι είναι και μία από τις πρώτες προτεραιότητες που αναφέρατε. Πράγματι εδώ είναι η χρονική στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδείξει ότι δεσμευόμαστε σε σχέση με την πολυμερή ημερήσια διάταξη και θέλουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερη παρατήρηση για δεύτερο ορόσημο. Η πολιτική για μια νέα ε, προσέγγιση στα εμπορικά θέματα. Είναι σημαντικό εσείς ως Προεδρία που θα λαμβάνετε από τις αποφάσεις για τις μελλοντικές προτεραιότητε να θέσετε τις προτεραιότητες σωστά. Και επανέρχομαι στον κατάλογο διαφόρων κρατών με τα οποία εμπλεκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και να πω ότι κάποιες από αυτές τις διαπραγματεύσεις διανύουν ήδη πολλά έτη ε, διαπραγματεύσεων υπό εξέλιξη και πρέπει να αξιολογήσουμε πού βρισκόμαστε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και μήπως να δούμε μήπως πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση ποια συνέχεια θα δώσουμε με χώρες όπως τη Mercosur ή το Συμβούλιο Συνεργασίας του Αραβικού Κόλπου για παράδειγμα Gulf Cooperation Council Σήμερα περισσότερο από ότι οποιαδήποτε στιγμή κατά το παρελθόν Πρέπει σε σχέση με τις φιλοδοξίε μα θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη στρατηγική μα για το εμπόριο. Με μια στρατηγική που θα ενδυναμώνει την εσωτερική ανταγωνιστικότητα των χωρών μα για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση και ανάπτυξη. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε στη ραχοκοκαλιά των οικονομιών μα που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, η ραχοκοκαλιά αυτή. Ερώτημά μου προ εμά. Πώ θα επικεντρωθείτε λοιπόν σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχεδιάζεται για παράδειγμα η στρατηγική πρόσβαση στην αγορά να αναδιαμορφωθεί ε, όσον αφορά τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να υπάρχει άμεσο feedback. Και δεύτερον, οι, σας, οι προτεραιότητες σας φυσικά έχουν ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανταποκρίνεται, αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους Ερώτησή μου, μπορεί κάτι να γίνει από κοινού όταν έχουμε το θέμα της οικονομικής διπλωματίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Helmut Scholz παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πραγματικά έχετε μια εκπληκτική ημερήσια διάταξη ως θεματολόγιο που παρουσιάσατε. Θέλω να πω προημίου ότι χαιρετίζω το θάρρος ε, λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα των θεμάτων της εμπορικής πολιτικής και στην εξωτερική δράση και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυθούν. Και εδώ αναφέρομαι στην ερώτηση πώς έχουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και πώς εσείς ως Προεδρία βλέπετε τα πράγματα. Μήπως υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ διμερών συμφωνιών και αυτού, αυτής της προσέγγισης τα αναφέρατε τα θέματα. Σε σχέση με την πολυμερή προσέγγιση δεν υπάρχει κάποια αντίφαση. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, να μας θεωρούν οι εταίροι ως εταίρους και να θεωρούμε και εμείς τους εταίρους ως εταίρους στον ΠΟΕ, θα πρέπει από κοινού με εκείνους να ρυθμίζουμε διατάξεις και προδιαγραφές για όλα αυτά τα θέματα. Δεν βλέπετε να υπάρχει εδώ ο κίνδυνος λόγω διμερών συμφωνιών αυτή η αρχή να υπονομεύεται. Διότι θα πρέπει να κατανοούν οι πολίτες γιατί ασκούμε το ένα ή άλλο είδος εμπορικής πολιτικής και φτάνουν στο θέμα της διαφάνειας. Δεν το κατανοώ και αναμένω από την Προεδρία του Συμβουλίου ένα σαφές μήνυμα σε σχέση με τα κράτη-μέλη η διαφάνεια <clears throat> μέσω, μέσω της ΟΝΣΙΤΡΑΛ ε, να μπορέσει να προχωρήσει με την προσυπογραφή της επιδιαιτησίας ε, στην οποία προχωρήσαμε. Έχουμε εδώ μία διαφορά μεταξύ αποστασιοποίηση λόγων και πράξεων. Εδώ θα είχε τη μεγάλη ευκαιρία η Λουξεμβουργιανή Προεδρία να κάνει το αποφασιστική σημασία βήμα για να σημειωθεί πρόοδο. Τρίτον, για το ISDS και τα συναφή θέματα του εμπορίου. Σύντομα, έχουμε τη νέα πρόταση τη Επιτρόπου για το εμπόριο Τραπέζης. Έχουμε τη στεναρή θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αναλάβει και πρωτοβουλία εδώ το, και, ε, το όργανο και το Κοινοβούλιο. Ποια είναι η θέση, για παράδειγμα, από πλευρά σας σε σχέση με το ISDS στις ε, διαπραγματεύσεις. Υποκλειστό πλαίσιο πρέπει να γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις ή μέσα σε ένα ανοιχτό πλαίσιο. Η Λουξεμβουριανή Προεδρία θα καταβάλει προσπάθειες έστω για το μικρό αυτό αποτέλεσμα όσον αφορά και το ψήφισμα της TTIP να γίνει αυτό το πρότυπο για την αξιολόγηση όλων των άλλων συναφών θεμάτων. Και το θέμα επίσης των επίμαχων ορυκτών και μετάλλων. Και ελπίζω ότι υπό την Προεδρία σας ε, γρήγορα θα καταλήξουμε σε μια επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών. Ευχαριστώ. Χέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη υπόθηκαν. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων όσον αφορά ε, τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις και την διαφάνεια. Και θα ήθελα να ρωτήσω τι συζητιέται μεταξύ των συναδέλφων σας σχετικά με το ISPS. Έχουμε αρκετά έγγραφα από διάφορα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν. Τα έγγραφα αυτά έχουν κάποια κοινά μεταξύ τους ε, και κάποιες διαφορές και υπάρχει μεγάλη αντίθεση απέναντι στο ISTS. Ε, Πώ συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση και όσον αφορά τα ορυκτά από τις εμπόλεμε ε, περιοχές θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση που θα κρατήσει το Συμβούλιο κατά τον τριμερή διάλογο και καθότι υπάρχουν ακόμα παρανοήσει σχετικά με τα ορυκτά από τις εμβόλεμες περιοχές. Ε, τι ακριβώς σημαίνει το να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ και κατά πόσο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να γίνει αρκετή ενημερωτική δουλειά από πλευρά της Προεδρίας, διότι θα είναι γελίο να έχουμε απέτηση για δέουσα επιμέλεια μόνο από τους ε, εισαγωγείς ε, και τους επεξεργαστές, ε, διότι αυτοί που ενδιαφέρονται ήδη κάνουν κάποια πράγματα. Χρειάζεται πιο φιλόδοξο επίπεδο, όπως άλλωστε έδειξε και η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου. Θα ήταν χρήσιμη λοιπόν η υποστήριξη της Προεδρίας σας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριος Μορέλη. Μορέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σταθώ μια στιγμή στο τελευταίο σημείο που ανέφερε ο υπουργό. Γιατί λόγω της ε, διάστασης του θέματος ε, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Ειδικά αν σκεφτούμε τις συνέπειες ε, στο μέλλον. Μιλάμε για τη σχέση με την Κίνα. Έτσι. Η Κίνα θέλει από το Δεκέμβριο 2016 να της αναγνωριστεί ε, ότι έχει οικονομία αγοράς. Με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ η Κίνα δεν ε, πληρεί καμία από τις προϋποθέσεις για να της δοθεί αυτό το στάτους. Έχει ξεκινήσει όμως μια έντονη διπλωματική εκστρατεία για να μετατοπίσει το θέμα από το τεχνικό επίπεδο στο πολιτικό επίπεδο. επίπεδο. Θέλω να σε επιστήσω την προσοχή Λουξεμβουργίας και Προεδρίας σε αυτό το γεγονός και να σας τονίσω κάποια σημαντικά στοιχεία. Το να δεχτούμε τη μετακίνηση της απόφασης σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από το τεχνικό στο τεχνικό, θα ήταν ένα πρόβλημα ε, νομοθετικό και θα αποτελούσε ένα επικίνδυνο ε, προηγούμενο. Εάν δεχτούμε αυτό το πράγμα αυτόματα, αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε μια βιομηχανική κρίση και συνεχεία μια κρίση στην αγορά εργασία σε διάφορες, ε, διάφορους τομείς της ε, ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σιδηρουργία, μηχανουργία κτλ. Και επίσης θα έπλητε και τους, ε, θα του και τους τίμιους, έτσι, τους νομότυπους εμπορικούς εταίρους μας. τελικά οι χώρες της Ευρώπης που είναι παραγωγή θα χάνουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω να το ξέρει αυτό η Προεδρία σας, ελπίζω να δράσετε με στεναρότητα αλλά και κυρίως ε, με διαφάνεια και για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Ευχαριστώ. Ε. Τέσσερις ομιλητές ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Θα θέλαμε όμως να δώσουμε τη δυνατότητα στον ε, ομιλητή να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το Λουξεμβούργο για την ανάληψη της Προεδρίας. Ελπίζω να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά της Λετωνίας, γιατί νομίζω ότι οι μικρές χώρες μπορούν να κάνουν την καλύτερη δουλειά. Δεν θα σας ρωτήσω σχετικά με το ISTS, όλοι σας ρώτησαν σχετικά με το θέμα αυτό, Απλώς θα ήθελα να πω ότι η ζωή συνεχίζεται. Οι συμφωνίες που συνάπτονται ήδη είναι ξεπερασμένες όταν έχουν υπογραφεί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι απλά η υπογραφή της συνθήκης. Και όσον αφορά την ΣΥΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά, θα ήθελα την, να ακούσω την ε, σαφή θέση της Προεδρίας, διότι ξέρουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις και ότι οι Καναδοί μας έχουν προσφέρει πολλά. Περιμένω λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία κατά τη διάρκεια ε, της Προεδρίας του Λουξεμβούργου και μάλιστα χωρίς αλλαγές, διότι αλλιώς μπορεί να υπονομευτούν οι εργασίες μας και επίσης ε, απαιτούνται ακόμα πολλά ε, στις σχέσεις μας με συνδεδεμένες χώρες όπως είναι η Νορβηγία και η Τουρκία. Και τέλος, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ακούμε μόνο, γράφουμε κιόλα. Έχω λοιπόν ένα προσωπικό δώρο προς τον φίλο μου, τον ε, Ζαν Ασελμπον. Λοιπόν, παρακαλώ. Η Μαρία έχει το λόγο. Merci. <laughs> <laughs> Ε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δεν θα σας συγχαρώ που λαμβάνετε, αναλαμβάνετε την ε, Προεδρία που παίρνετε τη σκητάλη. Ελπίζω να μπορώ να σας συγχαρώ όταν την παραδίδετε. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Καλή τύχη λοιπόν. Για δύο θέματα θέλω να μιλήσω κι εγώ και όπω είπε και ο David Μάρτιν θέλω να μιλήσω για τα μεταλλεύματα από τι περιοχές συγκρούσεων. Με ενδιαφέρει τα μάλλα αυτό το θέμα και χαίρομαι ότι θεωρείτε κι εσεί ότι είναι προτεραιότητά σα. Η τελευταία φράση σα με ανησύγησε λιγάκι όμω. Γιατί αφήνει να υπονοηθεί ότι υπάρχει ήδη έλλειψη κατανόηση για το τι αποφασίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Είμαι στη διάθεσή σα, ούτω ώστε να το ξανασυζητήσουμε αν χρειαστεί. Είπατε ένας κανονισμός δεν είναι καλός κανονισμός εάν έχει σαν στόχο να διώξει επενδυτές από τις χώρες όπου εκμεταλλευόμαστε αυτούς τους πόρους. Εμείς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε στον κανονισμό. Και όχι μόνο έχουμε θέση η οποία ε, αποφεύγει το να φύγουν οι επενδυτές, αλλά αποφεύγει και το να φύγουν οι επενδυτές από την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να βρούμε μια ισορροπία, λοιπόν, ανάμεσα τις επιπτώσεις που υπάρχει στις ε, τρίτες αυτές χώρες που υπάρχουν οι συγκρούσεις και τις επιπτώσεις που έχουμε εδώ στην ε, Ευρώπη, έτσι. Και είναι στη διάθεσή να το ξανασυζητήσουμε. Ένα άλλο θέμα, λεπτό και αυτό είναι, η ετικετοθεσία προϊόντων από απικίες. Θα γίνει νομίζω μια συνάντηση τον Οκτώβριο. Σκέφτεστε να προωθήσετε σαφή μέτρα ούτως ώστε να γίνει σεβαστό αυτό που αναγνωρίζετε σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή το θέμα των, ε, τι γίνεται με το θέμα των απικιών. Ευχαριστώ, Γιώργη Σούστερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα δύο θέματα. Καταρχάς η ΣΥΤΑ. Στο Κοινοβούλιο ε, έχουμε μιλήσει για την TTIP. Ε, πολλοί πιστεύουν ότι δεν δεν ε, θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη κανενός εάν ε, έχουμε τελείως διαφορετικές ε, συνθήκες για την ΣΥΤΑ από ό,τι για την TTIP. Θα υπάρξουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το ISTS κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και επίσης όσον αφορά την συμφωνία με την Ουκρανία. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό το ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Είναι σημαντικό να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να ε, καταστεί ότι η συμφωνία σύνδεσης ε, με την Ουκρανία δεν είναι συμφωνία κατά της Ρωσίας. Και ε, επίσης θα πρέπει να απαιτήσουμε μεταρρυθμίσεις από την Ουκρανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα η οικονομική συνεργασία να είναι προς όφελος ε, του πληθυσμού γενικότερα. Πώς ε, σκοπεύετε να συνεχίσετε στο θέμα της ε, Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα εκφράζω την ικανοποίησή μου για την λεπτομερή παρουσίασή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία, θα είναι επιτυχία όλων μας Κάνατε αναφορά στην αρχή σε κάτι που συμμερίζομαι απόλυτα σίγουρα στην πολιτική συνεκτικότητα. Θέλω να, απευθύνω έκκληση για την συνεκτικότητα της πολιτικής, ώστε αυτό το εξάμεινο να έχουμε τον εξυγχρονισμό των μέσων προστατευτικών μέσων εμπορίου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι με το TTIP διατηρήθηκε η, εχεμήθεια ή το απόρριτο. Υπήρξαν κάποια κράτη-μέλη που ήταν εναντίον της ε, διαφάνειας. Και έτσι πρέπει να ε, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε αν κάποιος είναι κατά να το γνωρίζουμε. Να μπορεί να υπάρξει όμως η διαφάνεια. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας ποια προτεραιότητα θα δίνατε σε σχέση με αυτό, σε σχέση με τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα. Αναφέρατε λεπτομερώς κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να ξέρουμε την Κούβα τι θα γίνει. Όσον αφορά τη Χιλή, Ποιο χρονοδιάγραμμα και χρονορίζοντα έχετε. Ποια προτεραιότητα δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον εξυγχρονισμό για τη συμφωνία με την Χιλή. Ένα θέμα ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Είναι σημαντικό προ αυτή την σκοπιμότητα το σκόπινγκ να έχει και την προοπτική τη ισότητα των φύλων στι πολιτικέ ε, και τη μελέτη επιπτώσεων. Και τέλος υπάρχει ένα θέμα που πολιτικά είναι περίπλοκο μένα αλλά είναι απόλυτα αναγκαίο Κάθε φορά όλο και απομακρυνόμαστε πιο πολύ από τους πολίτες και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα θα πρέπει να μας προβληματίσει. Πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση, ποια Ευρώπη επιθυμούμε. Είναι σημαντικό να εμπλακούν τα κράτη-μέλη στις αρχές και αξίες που υπερασπιζόμαστε εμείς στην Ευρώπη. Ως προς αυτό θα ήθελα να γνωρίζω αν μπορείτε κάτι να κάνετε για να ανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη σε σχέση με τις αρχές και αξίες της Ένωσης όσον αφορά τους πολίτες μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι περιμένει κανεί τώρα από τον Υπουργό κύριο Άσελμπορ να απαντήσει αναλυτικά σε όλες τι ερωτήσει. Αυτό είναι αδύνατο. Θα του δώσω αμέσω το λόγο και νομίζω θα δώσει κάποιε γενικές απαντήσει. εάν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε, μπορείτε να συνομιλήσετε διμερώς μαζί του από σεβασμό προς εσένα θα ε, μιλήσω τη δική σου γλώσσα. Ε, ε, να ξεκινήσω από το τέλος. Είμαι υπουργό Εξωτερικών και αυτό που κάνω εδώ είναι συμπληρωματική μου δουλειά, την οποία όμως γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα. Να ξεκινήσω από το τέλος, από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα από τα ποια φιλοσοφία αντιπροσωπεύουμε, είχε ένα καθήκον αυτό το Σαββατοκύριακο να εμποδίσει ένα Brexit. Αυτό θα ήταν μοιραίο, κατά τη γνώμη μου, για την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το Eurogroup, ε, αν η Ευρωζώνη θα είχε ε, επιβιώσει σε περίπτωση ενός Brexit. Χαίρομαι που τελικά οι δύο μεγαλύτερες και σημαντικότερες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία, συμφώνησαν. Και θα περάσω τώρα στην Κούβα. Γνωρίζετε ότι καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες. Η ύπατη εκπρόσωπος βρέθηκε στην Κούβα. Είναι σημαντική η χώρα αυτή. Ε, έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες και θα πρέπει να οικοδομήσουμε σχέσει ε, με τη χώρα αυτή, κάτι σημαντικό και για την Κούβα και για μας. Όσον αφορά τη διαφάνεια και το TTIP, μπορώ να επαναλάβω μόνο ότι είναι το α και το ω, διότι χωρί διαφάνεια το κοινοβούλιο σα δεν πρόκειται ποτέ να υπερψηφίσει την συμφωνία αυτή, ούτε άλλωστε πολλά εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω επί Ιταλικής Προεδρίας είχαμε συζήτηση στο Συμβούλιο όπου δεν τονίστηκε τόσο πολύ η διαφάνεια. Νομίζω όμως ότι τώρα πια ακόμα και στο Συμβούλιο δεν περιμένει κανείς ότι θα μπορέσουμε να εξαπατήσουμε κανέναν. Θα πρέπει να αποκαλύψουμε όλα τα στοιχεία. Και θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε και η Σεσίλια Μάλμστρομ θα πρέπει να πιέσουμε τους ε, Αμερικανούς, διότι χωρίς διαφάνεια δεν θα λειτουργήσει. Όσον αφορά την Ουκρανία, επισκέφθηκα τη χώρα πριν δύο εβδομάδες. Συνομίλησα με τον ε, πρόεδρο Ποροσέγκο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ουκρανίας και το λέω αυτό ως Υπουργός Εξωτερικών είναι ο καρκίνος της διαφθοράς Υπάρχει διαφορά παντού. Ήδη απολύθηκαν πολλοί δικαστές, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο εργάζεται σκληρά πάνω στη συνταγματική μεταρρύθμιση. Τον ε, Ιούλιο θα υποβληθεί ένα νέο σχέδιο με περισσότερη αυτονομία για τις περιφέρειες. Αυτό είναι θετικό και άλλο θετικό σημείο είναι ότι και για τις τοπικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο προβλέπεται μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Πιστεύω ότι η διαφορά στην Ουκρανία συνδέεται και με τα μονοπόλια. Όσο συνεχίσουν να υπάρχουν, τόσο θα υπάρχει μια ολιγαρχία την οποία θα πρέπει να καταπολεμήσουμε στη χώρα αυτή. Στην Ρήγα καταφέραμε να διατηρήσουμε τις ελπίδες για τις ε, τρεις ε, χώρες με συμφωνία σύνδεσης. Παρότι ήταν δύσκολες οι συνομιλίες, είμαι πεπισμένος ότι και η Προεδρία μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε οι τρεις χώρες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης ε, να μπορέσουν να συνομιλήσουν μαζί μας για το πώς να, μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα. Όσον αφορά την ε, συμφωνία ΣΥΤΑ, ε, η Προεδρία δεν μπορεί να προωθήσει το θέμα αυτό. Στα χέρια σας βρίσκεται λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Χωρίς τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε, να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα την συμφωνία αυτή. Έχετε λοιπόν αυτήν την πολύ σημαντική αρμοδιότητα. Δεν θέλω να εμπλεκώ σε διαφωνίες εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείε και εδώ ε, εστάλησαν τις τελευταίες μέρες σε σημαντικά μηνύματα. Έχουμε την αρχή TPA για την πρόθεση του εμπορίου. που ε, ασχολείται με όλες ε, τις εμπορικές ε, συμφωνίες και νομίζω ότι και εσείς στείλατε σαφές μήνυμα και είμαι πεπισμένος, μπορεί να κάνω λάθος, ότι πρόκειται για θετικά μηνύματα ώστε και το ISDS να μπει σε διαφορετικό δρόμο. εάν ε, μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ISDS νέας γενιάς και άκουσα ότι οι Καναδοί θα μπορούσαν ενδεχομένω να συζητήσουν το θέμα αυτό μαζί μας, τότε θα ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο Έξι χώρες ε, του Συμβουλίου, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, οι κάτω χώρες ε, και ε, εμείς έχουμε συνεργαστεί πάνω στο θέμα αυτό και νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν απέχει πολύ από κάτι τέτοιο. Μιλήσατε για μόνιμο δικαστήριο, όχι δικηγόρους, ανοιχτές διαπραγματεύσεις το Συμβούλιο, τουλάχιστον η δική μας Προεδρία, θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδιαφέρον είναι το θέμα της ετικετοθεσίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, καταβάλλονται εδώ και καιρό προσπάθειες ε, σχετικά με την ετικετοθεσία. Ως πρόεδρος ε, του Συμβουλίου ε, δεν είμαι αρμόδιος ε, για κάτι τέτοιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. Νομίζω ότι 17 ή 18 χώρες θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό. Η Φεντερίκα Μογκερίνη συνεχίσει τις προσπάθειες και κάνει τα απαραίτητα. Σωστό θα ήταν οι καταναλωτές να γνωρίζουν ε, όταν καταναλώνουν προϊόντα από κατεχόμενες περιοχές. Πιστεύω ότι η γραμμή που έχουμε διατηρήσει είναι αυτό που περιμένει κανείς από την Ευρώπη και ακολουθεί και το διεθνές δίκαιο. Θα με συγχωρήσετε που διατρέχω τόσο γρήγορα τα θέματα αυτά. Έχουμε ε, τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Πιστεύω ότι και στο Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό υπό την οπτική της ηθικής. Ε, ε, Έχουμε την περιοχή των μεγάλων λιμνών ε, στην Αφρική και ως Υπουργό Εξωτερικών πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε σαφή γραμμή στο θέμα αυτό. Γνωρίζουμε ε, για ορυκτά τα οποία γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτούν ε, τέτοιε. Ε, σειράξεις δεν μπορούμε να τα εισάγουμε στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν σωστή πιστοποίηση. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει για τον εξοπλισμό ε, βασανιστήριων ε, και για την ε, θανατική ποινή. Μιλήσαμε για τις κυρώσεις απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Όταν γνωρίζουμε ότι κάτι χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για το βασανισμό ανθρώπων ή για την εκτέλεση ανθρώπων, θα πρέπει να φροντίσουμε το Συμβούλιο να καταλήγει στις ε, σωστές αποφάσεις. Όσον αφορά την Κίνα, διστάζω να απαντήσω. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον της Ιταλίας και άλλων χωρών από τον βορρά της Ευρώπης που μπορεί να έχουν διαφορετική θέση, αλλά ε, Επί της αρχής η Κίνα είναι πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος για μας. Πριν δέκα χρόνια θα μπορούσα ήδη να σας είχα υπογράψει ότι ε, η Κίνα θα έχει αυτή τη θέση σε 10 χρόνια. Πρέπει να περιμένουμε την νομική ανάλυση για να δούμε σε τι συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Ε, όσον αφορά το ISTS απάντησα, όπως επίσης και για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Όσον αφορά την ε, σύμβαση του Μαυρικίου, έξι χώρες έχουν υπογράψει. Το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Ε, έχουν σκοπό να προσχωρήσουν και ελπίζω να το κάνουν αυτό και άλλες χώρες. Φτάνουμε στη διάσκεψη στο Ναϊρόμπι. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί, αλλά ως Προεδρεύων ε, έχω δεσμευτεί να επισκεφτώ τον Ναϊρόμπι. Χθες ε, συνομιλήσαμε την Σεσίλια Μάλμστρομ και είπαμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, το 90% της ε, ανάπτυξης ε, πραγματοποιείται εκτός Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά όλα τα θέματα που άπτονται του διεθνούς εμπορίου για την Ευρώπη. Πολλοί με έχουν ερωτήσει σχετικά με τις διμερείς και τις πολυμερείς σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι όσο είναι δυνατόν θα πρέπει να λύνουμε τα θέματα σε πολυμερές επίπεδο. Τι άλλο είχαμε. das war die erste Frage, die ersten Fragen von äh, Αυτά σε σχέση με τις πρώτες ερωτήσεις της κυρίας Ρέντινγκ. Συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις βέβαια που οδηγούν στο ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη προσέγγιση και σε σχέση με χώρες ε, που έχουν ανάγκη να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στην προσέγγιση μου ανέφερα τι συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα και το είδατε. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά. Φυσικά με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Και αν, και εγώ δεν είμαι μόνο υπέρ της συνέχειας και της συνεκτικότητας, είμαι και υπέρ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να υπάρξει και κάποια αναθεώρηση των πραγμάτων για τις χώρες BRICS Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, ε, Ρωσία θα πρέπει σε σχέση με αυτές να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ένα ε, διαφορετικό τρόπο. Έχουμε και εντολή σε σχέση με τη διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητεί κυρία Ρέντινγκ να διασφαλιστεί ότι με ιδιαίτερη προσοχή θα διεξαγάγει αυτές τις διαπραγματεύσεις η Επιτροπή και είμαι πεισμένος ότι το Συμβούλιο και όλοι θα παρακολουθήσουν με πολύ μεγάλη προσοχή και ε, εκ του σύνεγγης και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τα τέλη του έτους έχοντας πει ότι και το σημαντικότερο ήταν ότι σε αυτό το θέμα το πιο σημαντικό είναι ότι οι υπηρεσίες μας που μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταχτούν, να εντάσσουν τις προσπάθειές τους αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να μπορούν να, να δράσουν και σε σχέση με την TTIP συμφωνούμε απόλυτα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι τόσο διαφορετικές οι προσεγγίσεις ε, και κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουριανής Προεδρίας θα κάνουμε ότι περνά το χέρι μας, να σημειωθεί πρόοδος. Δεν θα τα καταφέρουμε όλα βέβαια και όλα να ε, με ένα μαγικό ραδί να τα ρυθμίσουμε αλλά όπου είναι ανάγκη να γίνει κάτι θα καταβάλουμε προσπάθειες η, η πόρτα μου είναι ανοιχτή για να, έχω, να μπορώ να παρακολουθήσω τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστούμε θερμά Υπουργέ. Σας Ήταν ευρύτατο το φάσμα των παρεμβάσεων αυτών και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. So, liebe Kolleginnen und Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε πολύ καλά και περνάμε στο σημείο 16 τώρα. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Πρόκειται για την συνεργασία με την Τουρκία στην Τελωνιακή Ένωση και την περαιτέρω εξέλιξη αυτής της συνεργασίας στις 12 Μαΐου η κυρία Μάνστρομ και ο Υπουργός Οικονομικών της ε, Τουρκίας ε, συζήτησαν πώς αυτή η τελωνιακή ένωση με την Τουρκία θα μπορέσει να εξυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί. Είναι 20 ετών, ε, έχει 20 έτη ηλικία και μια αναβάθμιση αυτής της συμφωνίας είναι κάτι σκόπιμο και πρέπει να γίνει. Κατά τούτο λοιπόν εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ενημέρωση για το έργο αυτής της ομάδας εργασίας για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας για την Τελωνιακή Ένωση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ένας παλαιός ε, γνωστός δεν είναι ε, πρεσβήτης αλλά ένας πολύ καλός γνωστός μας ο Ιγνάσιο Βεσέρο είναι παρόν που όχι <clears throat> ως κύριος διαπραγματευτής για την TTIP παρευρίσκεται σήμερα αλλά ως προεδρεύων σε αυτή την ομάδα εργασίας για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας για την Τελωνιακή Ένωση με την Τουρκία. Χαίρομαι Νάτσο που είσαι εδώ. Παρόλες τις διαπραγματεύσεις για την TTIP βρήκε τον χρόνο να μας εκθέσει τα σχετικά. Έχεις τον λόγο Ιγνάθιο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ και κάνω και ένα time out από τις διαπραγματεύσεις TTIP για να σα ε, εξηγήσω τι συζητήσει που έχουμε κάνει με την ε, Τουρκία για να εξυγχρονίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Το πρώτο που θέλω να πω είναι οικονομικό. Είναι ένα ε, σημαντικό εμπορικό εταίρο η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο έκτο σημαντικότερο εταίρο. Είναι το 4% του εμπορίου μα. Πέρα από τι πολιτικέ αποχρώσει των σχέσεών μα με την Τουρκία, από εμπορικής και οικονομικής σκοπιάς η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση του Επιτρόπου Δεχού το Φεβρουάριο του 2014 ε, να δημιουργήσει ε, μια ομάδα υψηλών, επιπέδων υψηλών ε, υπαλλήλων υψηλού επίπεδου για να εξυγχρονίσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία ήταν ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντική η Τουρκία. Δύο λόγοι ε, σε δύο λόγους εδράζεται αυτή η απόφαση. Να γίνει μια κοινή αξιολόγηση από την Τουρκία και την Κομισιόν ότι η Τελωνιακή Ένωση παρότι ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην, στο μετασχηματισμό της Τουρκίας και στην ε, στενότερη οικονομική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα και ήταν καιρός να το εξυγχρονίσουμε και να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Νομίζω ότι αυτό επίσης ότι από ευρωπαϊκής πλευράς υπήρχε μια έλλειψη ικανοποίηση, μια δυσαρέσκεια. Σε πολλές περιπτώσεις ε, η Τουρκία δεν ε, σεβόταν τις δεσμεύσεις της Θελωνιακής Ένωσης και δεν είχαμε ένα αποτελεσματικό ε, εργαλείο για να επιλύσουμε τα προβλήματα με Τουρκία με βάση τους θεσμούς που προβλέπει η Θελωνιακή Ένωση. Από τουρκικής πλευράς υπήρχε επίσης μια ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται όλο και περισσότερες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με σημαντικούς εταιρικού, ε, εμπορικούς εταίρους, ε, μερικοί πολύ σημαντικοί και ήταν δύσκολο να, κρατήσει, να κρατήσει την ισορροπία γιατί η ίδια η Τουρκία δεν διαπραγματεύεται τέτοιες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τις τρίτες αυτές χώρες. Δεύτερον, υπήρχε μια γενική αναγνώριση ότι η Τελωνιακή Ένωση που χρονολογείται εδώ και μια εικοσαετία έχει ξεπεραστεί για να λάβει υπόψη τα νέα στοιχεία της εμπορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πολλά στοιχεία των εμπορικών σχέσεων δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της ε, Τελωνιακής ε, Ένωσης. Με βάση αυτά τα δύο στοιχεία καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κάτσουμε μαζί με την Τουρκία για να αναλύσουμε πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε τις σχέσεις μας. Και γι' αυτό ε, ετοιμάσαμε την έκθεση που παρουσιάσαμε στους πολιτικούς ανωτέρους μας και η Επίτροπος Μάστρομ και, η και ο Τούρκος ομόλογός της ε, το επικύρωσαν. Ε, παρουσιάστηκε το Μάιο του 2015, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα σταθώ σε κάποια βασικά στοιχεία. Υπάρχει πρώτον η αναγνώριση ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότερο εργαλείο για να διευκολύνουμε τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου της Τουρκίας με τις χώρες που έχουν ήδη διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό μέλημα, σοβαρή ανησυχία της Τουρκίας και θέλουμε να ενισχύσουμε τους νομικούς μηχανισμούς ούτως ώστε να το καταστήσουμε αυτό δυνατό. Δεύτερον, συμφωνούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επίλυση των διαφορών στα πλαίσια της Τελωνιακής Ένωσης, ούτως ώστε να υπάρχουν ανησυχίες για τις δεσμεύσεις που δεν έχουν γίνει σεβαστέ από κάποιον εταίρο να έχουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για να επιλύονται αυτέ οι διαφορέ. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, για πρώτη φορά ε, συμφωνήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να διευρύνουμε τι εμπορικέ μα σχέσει για να καλύψουμε θέματα τα οποία δεν καλύπτει η Τελωνιακή Ένωση αλλά που είναι κρίσιμα ε, σε όλε τι ε, μοντέρνε εμπορικέ σχέσει. και συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται να αναπτύξουμε τι σχέσει μα για τι υπηρεσίε και για τις ε, κρατικές προμήθειες και για τη γεωργία, καθώς και τις, ε, τα θέματα των γεωγραφικών ενδείξεων και των ε, SPS, το, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων δηλαδή. Αυτά τα στοιχεία αναφέρει η έκθεση που επικυρώθηκε και από τις δύο πλευρές. Τώρα πρέπει να υπάρξει η επόμενη φάση. Θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αντικτύπου από την Κομισιόν και έχουμε πλησιάσει στη στιγμή εκκίνηση στη διαδικασία μελέτη αντικτύπου για να λύσουμε τις διάφορες επιλογές που έχουμε και να βελτιώσουμε τη σχέση μας με την Τουρκία. Και όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μελέτη αντικτύπου, τότε θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε μια πρόταση, στο, θα την υποβάλουμε στο Συμβούλιο, ε, για να λάβουμε διαπραγματευτική εντολή για να καλύψουμε αυτές τις νέες ε, σημαντικές ε, εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που έχουμε κάνει στις ε, σχέσεις μας με την Τουρκία. Είναι σημαντικό το ότι αποφασίσαμε τώρα να εξυγχρονίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις και αυτή θα είναι μία από τις σημαντικές μάλλον εμπορικές πρωτοβουλίες που θα πρέπει να προωθηθεί στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι εδώ στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχετε για την πρωτοβουλία αυτή. Αλλά η εισαγωγική μου παρέμβαση πρόεδρε θα σταματήσει εδώ. Ε, can you give us a timeline for... Μήπως θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη αντικτύπου και την εντολή. θα περιμέναμε να ξεκινήσει η μελέτη αντικτύπου ήδη τον Ιούλιο και αν όχι τότε αμέσως μετά τις Έλληνες διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και τότε θα παρουσιαστεί μια πρόταση εντολής στο Συμβούλιο. Δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος, σας δίνω ένα γενικό χρονοδιάγραμμα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πορέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρέμβω για την Τουρκία, που είναι στρατηγικό θέμα, στρατηγική χώρα για το μέλλον της ε, Ευρώπης και που παρακολουθώ πραγματικά από κοντά στο, στα πλαίσια του Monitoring Group. Τη ομάδα παρακολούθηση που για πρώτη φορά με αυτό το κοινοβούλιο δημιουργήθηκε. Σα ευχαριστώ επίσης Κομισιόν για την παρουσίασή σας. Η Τουρκία είναι στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο λόγω ιστορίας και λόγω πολιτικής, αλλά και λόγω γεωγραφίας φυσικά. Από τη Βυζαντινή περίοδο είχαμε, είχαμε την Ιερά Πύλη, όπου η Ιερά Πύλη πάντα έπαιξε έπαιζε η Τουρκία πάντα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, και με τη θρησκεία της και τα λοιπά. Η Τουρκία ε, δημιουργεί ε, αντίθετα αισθήματα εδώ στην Ευρώπη. Εδώ σε αυτό το βήμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λογικά. Η Τουρκία είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Εμείς πρέπει να ελεπιδράσουμε και από και η Άγκυρα ε, έχει μια οικονομία με εξελίξει και έχει πάρα πολλές διμερείς σχέσεις έντονες με διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε παγώσει την ε, διαδικασία ένταξης της Τουρκίας γιατί υπάρχει και έλλειψη ε, ενδιαφέροντος και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει μια διαφορία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε για τις εμπορικές πολιτικές μας που είναι αλεξαρτώμενες. Εδώ, και κυρίως σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέδειξε ένα δρόμο ε, μέσω της ε, Τελωνιακής Ένωσης, αλλά που δεν καλύπτει τις υπηρεσίες, τις ε, δημόσιες προμήθειες και τα γεωργικά. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις ε, συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες χώρες. Αυτό είναι ένα νέο δυναμικό που προσκρούει όμως σε μια νέα πραγματικότητα όπως πρόκειψε από την ε, προβληματισμό της Monitoring Ε, ο Λουκ Τεβίν της Γενικής Διεύθυνσης ε, Trade μας είπε την τελευταία φορά ε, ποια είναι η κατάσταση στο πακέτο διαπραγματεύσεων που είναι απαραίτητο για να καταλάβουμε και τα διάφορα κρίσιμα σημεία. Παραδείγματος χάρη το γενικός ότι δεν, χάρη δεν υπάρχει μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Ακούσαμε επίσης διάφορους Ευρωπαίους stakeholders σε σημαντικούς τομείς, κλωστεφαντουργικά και τα ε, τα είδη άθλησης, ε, φαρμακευτικά, υπηρεσίες, τεχνολογίες, ε, πληροφορικής και αλκοολούχα ποτά. Ε, εδώ έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν, υπάρχει διακριτική μεταχείριση από τους Τούρκους. Ε, αυξάνουν δυσανάλογα τα, τους δασμούς και βάζουν και μη τελωνιακούς, ε, μη θεσμολογικούς συγγνώμη θρασμούς ε, δυσανάλογους. Επίσης κάνουν τυχαίους ελέγχους ε, πριν ήταν στο 5-10%. Ενώ τώρα έχουν φτάσει στο 60-70% με τελώς αυθαίρετο τρόπο. Ζητάνε επιπλέον ε, παρα, ε, πληροφορίες για ευαίσθητα δεδομένα. Και έχουν βάλει και νέοι θασμοί από 25 έως 50% σε διάφορα είδη, μεταξύ των οποίων και τα υποδήματα. Αυτοί οι δασμοί, οι περαιτέρω δασμοί, δεν αφορούν προϊόντα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο ε, προϊόντα τρίτων χωρών. Αυτό έχει επιπτώσεις παρόλα αυτά σε Ευρωπαίους διανομής ε, προϊόντων μη ευρωπαϊκών, έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα, να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση και πολύ συγκεκριμένη, ούτως ώστε και να διευρύνουμε τις σχέσεις μας, ε, τις οικονομικές ε, και τις διμερείς με την Τουρκία, αλλά και να σταματήσουν αυτές οι διακριτικές πρακτικές που παρατηρήσαμε τελευταίως. Ε, η Τελωνιακή Ένωση είναι πολύ παλιά, πρέπει να ανανεωθεί και για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Οι Τούρκοι ε, φαίνονται πολύ ενοχλημένοι. Υπάρχει νομίζω διεύρυνση για, υπάρχει περιθώριο για διεύρυνση των εμπορικών ροών μας. Ε, υπάρχει ενόχληση από μέρους των Τούρκων γιατί κάνουν τις τι TTIP. Κάνουν επιλογές αντιεμπορικές ας πούμε, ε, μέσω δασμών και μέσω άλλων μη δασμολογικών φραγμών. Ε, νομίζω ότι το Monitoring Group μπορεί να προωθήσει τον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ των μελών της Επιτροπής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τουρκικές αρχές που είναι υπεύθυνε για την, ε, την διαδικασία εξυγχρονισμού, ε, οι εμπορευόμενοι της Ευρώπης και της Τουρκίας, νομίζω ότι άμα συζητήσουμε θα μπορούμε να, έχουμε, να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, να σας πω κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίσουμε στο Monitoring Group. Καταρχάς τα πιο πολιτικά θέματα αφορούν τις νέες σχέσεις, ε, τις νέες δυναμικές που προκύπτουν στον πολιτικό χάρτη της Τουρκίας. Μπορεί να, οι πολιτικές αυτές επιλογές μπορεί να επηρεάσουν τις διμερείς σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμπορικά θέματα και σε ό,τι αφορά την ενεργειακό ανεφοδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια. Η Κομισιόν τι μπορεί να κάνει, ε, γιατί υπάρχει μια στρέβλωση στην Τελωνιακή Ένωση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρακτικές που είναι πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης ουσιαστικά. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα να στήσω το λόγο. Νομίζω ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην επαναξιολόγηση των εμπορικών μας σχέσεων με την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία πρόσφατα έγιναν κοινοβουλευτικές εκλογές και ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση και μάλιστα προς μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία. Ταυτόχρονα, συνάπτοντας μια σειρά εμπορικών συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και άλλες χώρες, αυτό επηρεάζει και το εμπόριο μας με την Τουρκία. Και έχουμε εδώ δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, βλέπουμε και ακούμε πολλά παράπονα αλλά και ενθάρρυνση από πλευράς Ευρωπαίων επιχειρηματιών να κάνουν κάτι διαφορετικό. Οι προηγούμενες μας συμφωνίες με την Τουρκία είναι προφανώς τώρα πια απεκολιωμένες. Ακούμε όμως και θεμητές απαιτήσει και παράπονα από την τουρκική πλευρά. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση και από τις δύο πλευρές και να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Διότι είναι καλό πράγμα οι εμπορικές συμφωνίες εφόσον είναι προς αμοιβαίο όφελος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βρίσκεται και σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Τάντη. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπερσέρο για την παρέμβαση και την ενημέρωση και τον κύριο Μπορέλη. για την παρουσίαση της εργασίας που γίνεται στο Monitoring Group, στην ομάδα παρακολούθησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά, το είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, λόγω της σημασία που έχει η Τουρκία. Λόγω όγκου, ε, λόγω εμπορικών σχέσεων, λόγω εξαγωγών και εισαγωγών στην Ευρώπη. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η ενημέρωση. Η Τουρκία έχει μία συνθήκη που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να ανανεωθεί, να επικαιροποιηθεί. Είναι ανάγκη αυτό. Και το έχει συνειδητοποιήσει και η Ευρώπη και η Τουρκία. Υπάρχουν επίσης άλλοι τα πολιτικά θέματα, γιατί η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, που αφορά την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Είναι ένα σημαντικότατο εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας, το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να επιληθεί ε, στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Πέρα όμως από αυτό το πολιτικό στοιχείο, είναι σαφές ότι εμείς θα πρέπει, και γι' αυτό γίνεται νομίζω και η σημερινή συνεδρίαση, και χαίρομαι που διαπραγματευτής ο κ. Μπερσέρο είπε ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να γίνει να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ασχοληθούμε με αυτή τη νέα συνθήκη που θα πρέπει να συνάψουμε με την Τουρκία. Εξού και η πίεση για νέε διαπραγματεύσει κτλ. Δεν έχουμε λησμονήσει καθόλου τη σημασία του θέματο λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ειδικά τι υπηρεσίε, του δημόσιου διαγωνισμού και προμήθειε. Αυτά μα ενδιαφέρουν και εμάς τα θέματα, αλλά και την Τουρκία. Από πλευρά μα λοιπόν, απόλυτη υποστήριξη, για να ζητήσουμε πολύ γρήγορα αυτή την, να, να γίνει καταρχάς η μελέτη αντικτύπου, η οποία έχει προβλεφθεί όλα αλλά να ολοκληρωθεί όλα αλλά το συντομότερο δυνατόν να, στείλει μια, να δώσει μια εντολή στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να συσφίξουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με την Τουρκία, να έχουμε μια συνθήκη πιο μοντέρνα που θα εντάσσεται στα πλαίσια των εμπορικών εξελίξεων και των διαπραγματεύσεων που κάνει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Äh, ναι, το ECR συμφωνεί με την έκθεση του εισηγητή και με την Κομισιόν αναφέρονται τα σημαντικά προβλήματα. Η παρούσα κατάσταση της Τελωνιακής Ένωσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία δεν είναι ικανοποιητική ούτε για τη μία πλευρά ούτε για την άλλη. Η Τουρκία παραπονιέται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει συμφωνίες εμπορίου χωρίς να συμμετέχει η Τουρκία. και υπόθηκε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες ε, από την άλλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένα μέσα ε, σε περίπτωση προβλημάτων από πλευρά τη Τουρκία. Δηλαδή, λείπει ένα ικανοποιητικό μηχανισμό διαιτησία. Πιστεύω λοιπόν ότι για τους λόγους αυτούς θα είναι ωφέλιμη μια νέα σύγχρονη ε, συμφωνία με την Τουρκία που να περιλαμβάνει και τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτή είναι η θέση του ECR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μαρέικε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ιγνάσιο για την ενημέρωσή σου. Η Τελωνιακή Ένωση ήταν ένα βήμα προς την ε, προσχώρηση. Έχουν αλλάξει οι καιροί. Ο καθένας ε, έχει τις απόψεις του σχετικά με το αν αυτό είναι καλό ή όχι, αλλά εμείς θα θέλαμε να είχαμε δει περισσότερη πρόοδο. Ετούτη τη στιγμή ως αποτέλεσμα της έλλειψης πρόοδου ακούω όταν μιλώ με Τούρκους πολιτικούς πολλά παράπονα όσον αφορά τη λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σωστό να υπάρξει επικαιροποίηση. Ίσως θα ήταν χρήσιμο όμως να έχουμε και τη δική μας ε, αξιολόγηση όσον αφορά την επιτυχία της Τελωνιακής Ένωσης, διότι εγώ πιστεύω ότι ήταν ε, ωφέλιμη και για τις ε, δύο πλευρές. Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη στην μελέτη αντικτύπου, να έχουμε επαρκή στοιχεία και να μην βλέπουμε το θέμα μόνο από πολιτικής πλευράς. Δεδομένου ότι πολλά θέματα πολιτικοποιούνται στην Τουρκία και ότι υπάρχει μεγάλη υπόλωση, δυστυχώς, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της Τουρκίας. Γίνεται λόγος για νέες εκλογές για ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να συνεχιστεί η όλη διαδικασία και θα ήθελα να ρωτήσω ε, αν γνωρίζουμε τι περιμένει η Τουρκία και ποια είναι η πολιτική δυναμική, ε, αν δηλαδή πρόκειται να συναντήσουμε δυσκολίες. Πρόεδρος. Ναι, πράγματι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Πράγματι πιστεύω ότι η τουρκική πλευρά έχει δικαιολογημένα παραπονιέται όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν υπάρξει στην Τελωνιακή Ένωση. Θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, ποιοι είναι οι στόχοι της Κομισιόν όσον αφορά τη συμπερίληψη ρήτρα για την Τουρκία στις ε, συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η επικαιροποίηση της ε, Τελωνιακής Ένωσης θα διαρκέσει αρκετό καιρό και αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται υπό εκπόνηση πολλές σημαντικές συμφωνίες εμπορίου. Επίσης, όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημόσιες συμβάσεις, σε τι βαθμό θα ενσωματωθούν αυτά ε, στην ε, Νέα Τελωνιακή Ένωση. Δηλαδή η Τουρκία θα ε, είναι ουσιαστικό μέρος της ενιαίας αγοράς ή όχι ακριβώς. Και αναφερθήκατε στον τομέα των υπηρεσιών. Εάν κοιτάξουμε τις συμφωνίες ΤΙΖΑ, διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμφωνούν πάντα όσον αφορά τι υπηρεσίε, Πού βλέπετε λοιπόν να υπάρχει κοινό τόπο στον τομέα των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μαυρίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω να σημειώσω αρκετά πράγματα, γι' αυτό θα είμαι σύντομο Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι οι καλές ε, εμπορικές συμφωνίες δεν είναι απλά καλές, είναι εξαιρετικές εφόσον σέβονται το κράτος δικαίου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας εμπορικός κανόνας που να, ε, να θεωρείται ότι υπερτερεί το, τον, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας ε, λοιπόν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του εφόσον αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με το κράτος δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, του του λεχτέντος θα ήθελα να θυμίσω σε όλους ότι η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει την Τελωνιακή Ένωση απέναντι στην ε, Δημοκρατία της Κύπρου και ουσιαστικά μπλοκάρει οποιοδήποτε εμπόριο με την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, διάβασα μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία αναφέρεται εδώ αρκετές φορές, ε, δεν είναι όμως απόλυτα ισορροπημένη, δεν αναφέρεται στις απώλειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Κύπρου από το εμπάργο που εφαρμόζει η Κύπρος απέναντι στην Δημοκρατία της, της Κύπρου και άρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη παρατήρηση. Όσον αφορά τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, διαβάζω ε, από την έκθεση σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Νομικά δεσμευτική ρήτρα που να επιτρέπει στην Τουρκία να ε, ε, αποφελείται από τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Νομικά δεσμευτική ρήτρα, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν τα κράτη-μέλη μπορούν μόνο τους να αποφασίσουν και να μην δεσμεύονται από μια τέτοια συμφωνία. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι η εξής. Ε, είμαι υποστηρικτής του εμπορίου και θυμάμαι πριν μερικούς μήνες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου συζητήσαμε μία έκθεση σχετικά με την κακή συμπεριφορά της Βοσνίας Ερζεγοβίνης απέναντι στην Κροατία η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν σεβάστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν ε, σεβάστηκε την προτιμησιακή συμφωνία με την Κροατία. Και λάβαμε κάποια μέτρα στην περίπτωση αυτή. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο με την Τουρκία. Τόσο απλό είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι είναι θετικό να επικεντρωθούμε στην Τουρκία. Είναι πολύ μεγάλη χώρα ε, και ε, άμεσος γείτονας. Και ε, είναι πολύ καλύτερο που ακούμε για μια χώρα που θέλει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να ακούμε για τις χώρες που θέλουν να αποχωρήσουν. Η Τουρκία είναι ο έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας. Και τώρα με την κατάσταση στην Ουκρανία και με τη Ρωσία ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, προμήθεια ενέργειας. Ε, θα πρέπει να την διατηρήσουμε και να τη διαφοροποιήσουμε. Και η Τουρκία έχει εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και ανοιχτοί απέναντι στην Τουρκία, να συζητήσουμε θέματα ενδιαφέροντό μα και είμαι βέβαιο ότι και εκείνοι θα έχουν κάποιε ανησυχίε ή κάποιε σκέψει σχετικά με τον τρόπο που τους έχουμε αντιμετωπίσει εμείς. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το ελεύθερο εμπόριο. Καθότι η Τουρκία είναι χώρα τόσο κοντινή σε μας, όσο πιο σύντομα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα και να καταλήξουμε σε λύσεις, τόσο το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η σου δίνω το λόγο για να απαντήσεις. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους μίλησαν προς υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. Η σχέση με την Τουρκία έχει μια ισχυρή οικονομική και πολιτική συνιστόσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά ανησυχεί για την έλλειψη εφαρμογής από την Τουρκία βασικών υποχρεώσεων ε, υπό τη Συμφωνία της Άγκυρας και ελπίζουμε όταν φτάσει η στιγμή να αποφασίσουμε για την κίνηση των νέων διαπραγματεύσεων και την έναρξη των νέων διαπραγματεύσεων θα έχουμε μια κατάσταση που θα μας βοηθήσει για να επιλύσουμε το πρόβλημα που έχουμε με τη Συμφωνία της Άγκυρας. Τώρα, ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο στην Τουρκία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά η τουρκική κυβέρνηση έχει την άποψη ότι ανεξάρτητα από την πρόοδο στη διαδικασία ένταξης υπάρχει οικονομικό συμφέρον ε, για να ενισχύσει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη. Επί χρόνια δεν μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε διμερώς με την Τουρκία για θέματα όπως οι υπηρεσίες, ή κρατικές προμήθειες, γιατί μας έλεγαν ότι αυτά είναι κεφάλαια που ανήκουν στη διαδικασία διεύρυνση και θα αντιμετωπιστούν μόνο στα πλαίσια της διεύρυνσης. Ε, επομένως, αυτή η μετακίνηση ε, τη σημερινή τουρκική κυβέρνηση ήταν πολύ σημαντική. Αποφάσισαν ότι οι εμπορικέ σχέσει με την Ευρώπη είναι τόσο σημαντικέ που ανεξάρτητα από τι τροπή θα πάρει η διαδικασία ένταξη, υπάρχει λόγο να ενισχύσουν τι σχέσει αυτέ. Και αυτή ήταν μία ε, πολιτική απόφαση που πήρε η κυβέρνηση ΑΚΑΠΕ. Και την ε, συμμερίζονται και οι περισσότερες πολιτικές ε, δυνάμεις στην Τουρκία. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν προσέγγιση σε περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση στην Τουρκία. Από όλε τι ένδειξει και τα μηνύματα που μα στέλνει η Τουρκία, είναι, μπορούμε να πούμε ότι θέλουν πραγματικά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού της Τελωνιακής Ένωσης. Φυσικά είναι διαδικασίε του είπαμε που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου σωστή. Πρέπει να λάβουμε μια εντολή από το Συμβούλιο. Ε, υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να γίνουν πριν μπούμε σε διαπραγματεύσει με του Τούρκου. Αλλά από όλε τι ενδείξει που έχουμε από την τουρκική πλευρά φαίνεται ότι υπάρχει μια επιθυμία και μια διάθεση και ανοιχτό πνεύμα για να ξεκινήσει η διαδικασία εξυγχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης το συντομότερο δυνατό. Να μην σας ε, κλείσω και έναν άλλο βασικό παράγοντα στην τουρκική θέση. Είναι ότι ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτείες. Ε, η TTIP είναι η πιο μεγάλη εμπορική συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι στιγμής και για την Τουρκία θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εάν συνάψουμε μια εμπορική συμφωνία με ένα τέτοιο σημαντικό ε, εμπορικό εταίρο, ε, όπω είπα, χωρί η Τουρκία να έχει τη δυνατότητα να έχει σχέση ελευθέρω εμπορίου με τη ΣΥΠΑ, αυτό θα ήταν πρόβλημα για την Τουρκία. Αυτό έπαιξε ρόλο λοιπόν και έτσι εμείς ε, κρατούσαμε πάντα ενήμερη την Τουρκία για τις συζητήσεις που είχαμε στη ΣΥΠΑ και εξηγήσαμε στη ΣΥΠΑ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε ένα τρόπο ε, επίλυσης του θέματος ε, για τις σχέσεις ελευθέρου εμπορίου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Τουρκία. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά όποτε διαπραγματεύεται συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τρίτες χώρες και ειδικά με την Τουρκία και την Τελωνιακή Ένωση πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να ανοίξουν όταν ε, διαπραγματευόμαστε λοιπόν ε, συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες όπως την Κορία όταν ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις τους λέγαμε ότι πρέπει να συζητήσουν και με την Τουρκία και το πετύχαμε και τώρα η Κορέα με την Τουρκία έχει συμφωνία ε, ελευθέρου εμπορίου. Σε άλλες περιπτώσεις δεν, καταφέρουμε να πείσουμε, δεν καταφέρουμε να πείσουμε τις χώρες αυτές ε, τόσο εύκολα. Αλλά έχουμε μιλήσει και με τον Καναδά και με την Ιαπωνία για να ξεκινήσουν συζητήσεις ελευθέρου εμπορίου με την Τουρκία. Βεβαίως είναι στη θέλησή τους, έτσι, στη διακριτική του ευχέρεια. Εμείς επιμένουμε ότι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού της Θελωνιακής Ένωσης πρέπει να έχουμε μια ισχυρότερη δέσμευση ούτως ώστε να πείσουμε και τις τρίτες χώρες να θελήσουν να διαπραγματευτούν με την ε, Τουρκία. Μέχρι εκεί όμως μπορούμε να πάμε σε αυτό το πολύ περίπλοκο θέμα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη διαδικασία και αυτό θα πρέπει να το δούμε, αυτό το θέμα δηλαδή με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να το δούμε και στη μελέτη αντικτύπου. Και πρέπει βεβαίω να λάβουμε και τη σωστή διαπραγματευτική εντολή. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι δεν πρέπει σε όλη αυτή την προσπάθεια να χάσουμε και την εμπορική μα αυτονομία για το πότε θα ανοίγουμε και θα τελειώνουμε τη διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε. Απλώ θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρότερα κίνητρα για τρίτε χώρε, ούτω ώστε να αναπτύξουν τέτοιου τύπου εμπορικέ σχέσει και με την Τουρκία. Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη. Προφανώ ένα θέμα που πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν το αναφέραμε ρητά σε αυτά τα πλαίσια της ε, ομάδας υπαλλήλων υψηλού επίπεδου, αλλά θα είναι τμήμα ε, των νέων εταιρικών μας, ε, εμπορικών μας σχέσεων με την Τουρκία. Ε, κρατικές προμήθειες προφανώς είναι από τα θέματα. Ε, έχει εντοπιστεί και στην ομάδα εργασίας και στην έκθεση που έχει στην ομάδα εργασίας των ανώτερων υπαλλήλων. Είναι δύσκολο θέμα. Γιατί μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει ανοίξει αυτή την αγορά της σε τρίτες χώρες των κρατικών προμηθειών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει η Τουρκία να προσαρμόσει την νομοθεσία της ούτω ώστε να ευθυγραμμιστεί με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κρατικέ προμηθειέ. Ναι, δέχτηκαν με αυτό το θέμα τμήμα των διαπραγματεύσεων, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα είναι από τα δύσκολα, από τα ακαθόδη θέματα στι διαπραγματεύσει. Τι είδου ε, μηχανισμό επίλυση διαφορών, φυσικά και αυτό θα πρέπει να το δούμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα μοντέρνο ας πούμε, μηχανισμό ε, που έχουμε στις συμφωνίες ε, Ελευθερομπορίου. δηλαδή ε, νομικά δεσμευτικό μηχανισμό διαιτησίας, αντίστοιχο με αυτό που έχουμε στον ΠΟΕ και που μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το ζητήσει οποιοδήποτε από τα δύο μέρη. Ενώ στο μηχανισμό επίλυση διαφορών που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Τελωνιακή Ένωση πρέπει να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη. Όχι να το ζητήσει το ένα ή το άλλο είδαμε πόσα πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν οι επιχειρήσει μα ε, για τα μέτρα πούμε, που φυλάβει η Τουρκία, τα οποία είναι προφανώ σε κατάφορη παράβαση τη ε, συμφωνία. Και υπάρχουν ας πούμε, επιπλέον δασμοί ε, που επιβάλλονται ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση τη συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμή δεν είχαμε τον κατάλληλο μηχανισμό για να πολεμήσουμε ας πούμε, και να βρούμε τη λύση. Πρέπει να σα πω ότι δεν σκοπεύουμε να συνεχίσουμε Έτσι, ε, πρέπει να κάνουμε και διαβήματα σε πολιτικό επίπεδο για να σεβαστεί η Τουρκία τις δεσμεύσεις της και η Επίτροπος Μάτσομ ε, σε πάνω από μία περιπτώσεις έχει διαβιβάσει αυτό το μήνυμα στις τουρκικές ε, αρχές, τους τουρκικούς ομολόγους τους. Οι υπηρεσίε θα είναι δύσκολο θέμα. Θα υπάρξουν θέματα όπου η Τουρκία θα πιέσει στις διαπραγματεύσεις και θα ανεβέσει κάποια θέματα οι χερσαίε μεταφορέ, α πούμε, το αναφέρατε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα, ανησυχεί η Τουρκία και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, ζήτημα, αλλά σε κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ανταποκρίνεται στα αμοιβαία συμφέροντα για να θεωρήσουμε ότι η διαπραγμάτευση είναι επιτυχής. Δεν θέλω να σα δώσω την εντύπωση ότι θα είναι εύκολη διαπραγμάτευση, θα είναι περίπλοκη. Αλλά πιστεύουμε, όπως είπα και στην αρχή, ότι είναι η Τουρκία ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρου και πρέπει να έχουμε μια εμπορική πολιτική που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις σχέσεις μας. Ε, πρέπει να είναι και μοντέρνα και αποτελεσματική. Ευχαριστώ Ιγνάσιο και καλή τύχη βεβαίω στι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία αλλά και στι διαπραγματεύσει με τις ΗΠΑ ε, Πολιτείες για το TTIP. Ευχαριστώ. Τελειώνουμε τώρα αυτό το σημείο. Και πάμε στο σημείο 17 για τον προϋπολογισμό. Και έχουμε και τη γνωμοδότησή μας γι' αυτό. Απαρουσιάστηκε στις 27 Μαΐου το, ο προϋπολογισμός και υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και τώρα πρέπει να παρουσιάσουμε εμείς ε, την πρότασή μας για τον ε, προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ο κύριο Μπέγκε. Ο, ο μας ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Πράγματι, η δική μας δουλειά είναι τώρα να υποβάλουμε προτάσεις, να διατυπώσουμε τροπολογίες και θέλω να εκφράσω την, επιθυμ, την ελπίδα μετά από τη διαδικασία πέρσι που είχαμε να καταφέρει η Λουξεμβριανή Προεδρία να βρει μια καλύτερη οδό για τις διαπραγματεύσεις ε, από ό,τι κατά το παρελθόν διότι όσον αφορά τα πεπραγμένα κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο και όταν στις 8 και 13, 8 και 17 επιτυγχανόταν μια επίλυση ε, τότε θα πρέπει να είμαστε στο μέλλον πιο αποτελεσματικοί επιτέλους αλλά πραγματικά <clears throat> είναι στα χέρια του Συμβουλίου για να γίνει κάτι τέτοιο και παράλληλα με τη συνεδρίασή μας εδώ Έχουμε μια διοργανική ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο που ε, αυτή τη στιγμή συνεδριάζει όπου το πρόβλημα των ε, κρεμουσών πληρωμών, των πληρωμών από πλευράς ε, του προϋπολογισμού εξετάζει, ώστε το Συμβούλιο έχοντας συνειδητοποιήσει το θέμα προσπαθεί μερικά να βρει κομμάτι-κομμάτι τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Το λέω αυτό εκ προημίου, διότι στην αρχή, διότι όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου και ιδιαίτερα λαμβάνοντας ε, υπόψη το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα στην κατηγορία 4, το περιθώριο είναι πάρα πολύ περιορισμένο και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ περιορισμένο και το θέμα του τι θα απορρεύσει κατά το μέλλον όσον αφορά απαιτήσει, όσον αφορά τον προϋπολογισμό είναι κάτι το οποίο μένει μετέωρο και παραμένει σε εκκρεμότητα και πρέπει να αποφασιστεί. Έχουμε το σχέδιο τώρα ενώπιον μας για την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Σε πέντε σημεία προσπάθησα να συνοψίσω τα πράγματα. Αφενός εμένουμε και επιμένουμε να έχουμε μια επακή μια επαρκή πρικοδότηση με κονδύλια εκεί όπου είναι αναγκαίο και πραγματικά με φιλόδοξο τρόπο θέλουμε να δώσουμε συνέχεια αλλά στην υλοποίηση και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις συμφωνιών εμπορίου να τις δούμε σε μεγαλύτερο βάθος, να εποπτεύσουμε και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν, ίσως κάποια πράγματα να τροποποιηθούν. Είδαμε δεύτερον σε πολλές χώρες πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμιοποίηση την θεωρούν κάτι που συνδέεται άμεσα με απώλεια θέσεων απασχόλησης και με προβλήματα ύφεση. Και εδώ υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η επικοινωνία, ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία και πληροφόρηση από πλευρά τη Επιτροπή προς όφελος των πολιτών. Χρειαζόμαστε αυτή τη δουλειά για την επικοινωνία ώστε να διεξαχθεί μια ανοιχτή συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα με τους πολίτες. Ευτυχώς εδώ ε, στην ε, δική μας Επιτροπή έχουμε και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και την μελέτη που το κονδύλιο που αφορά μελέτες Πρέπει να δούμε ποια είναι η επιρροή των, μικρο... Ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων στην πολιτική αυτή και πώς μπορούν αυτές να διαδραματίσουν ένα ρόλο. Και να, να δούμε ότι υπάρχει μια ελαφρά αύξηση ως 2,2 στις υποχρεώσεις, 7,3 ε, στις ε, πληρωμές και εδώ τίθεται νομιμοποιημένα το ερώτημα σε σχέση με τους εταίρους αν είναι δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να επαρκέσουμε και να σκεφτείτε υπόψη για παράδειγμα τα προγράμματα υποστήριξης για την Ουκρανία και τις ανάγκες στην Ουκρανία για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη στις, ε, στα κονδύλια για την υποστήριξη, όλοι εμένουμε και επιμένουμε να υπάρξει υποστήριξη των αναπτυσσομένων κρατών, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση της ενδέκατης Υπουργικής Διάσκεψης ε, ε, για τα θέματα αυτά. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα σήμερα, θα παρακαλούσα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να απαντήσει, διότι έχουμε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση ήδη τον, την Παρασκευή λήγουν οι προθεσμίες. Και σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας του 2015 βλέπουμε αφενός 4,8 εκατομμύρια δεσμεύσεις υποχρεώσεων, 9,3 εκατομμύρια πιστώσεις πληρωμών και βλέπουμε για το 2016 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο 4,5 εκατομμύρια προβλέπουν για το κονδύλιο ε, για το εμπόριο Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια διακύμαση στις πιστώσεις πληρωμών. Σημαντικές ε, κιόλα διακυμάνσεις ε, ή έχουμε και ίσως και διπλασιασμό ή και πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ με τα πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα και πλαίσια. Θα ήθελα να έχω περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, διότι φυσικά έχει τη σπουδαιότητά του το θέμα για το ζήτημα ποιες τροπολογίες θα επιλέξουμε όσον αφορά τα επιμέρους κονδύλια. Όσον αφορά το σημείο 5 και ιδιαίτερα το θέμα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των business centers, πράγμα το οποίο μας απασχόλησε πέρυσι, θα ήθελα να επισημάνω εδώ κάτι. Έχω ακούσει κάποιες, κάποιες φήμες ή κάποιες ε, πληροφορίες ε, εν παρόδο που όμως δεν είναι καθοριστικές για το τι θα γίνει και θέλω να γνωρίζω πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν κάποιες, κάποια νέα στοιχεία, κάποιες πληροφορίες που δεν έχω ακόμα στη διάθεσή μου. Πρέπει να αναμείνω να δω τι θα απορρεύσει από αυτό το θέμα. Παρότι βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες και το κείμενο έτσι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, να ενημερωθεί για να είναι επίκαιρο. Όσον αφορά το θέμα των τροπολογιών στη συνέχεια για το σχέδιο προϋπολογισμού θα έλεγα ότι μπορούμε να προτείνουμε και να ε, καταθέσουμε τροπολογίες σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα ζητήματα αυτά έναντι της πρότασης του Συμβουλίου. Δεύτερον, το ζήτημα αυτής της μελέτης ε, για τον διοικητικό προϋπολογισμό να υπάρξει κάποια αύξηση σχετικά και κατά τα άλλα θα ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στου κύριους συζητητέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή για τη δουλειά που ήταν πολύ πλήρη, πολύ δύσκολη για να συντάξει αυτή την, αυτό το κείμενο για τον προπολογισμό. Κάθε φορά είναι τόσο δύσκολο. Να σκεφτούμε το εξή και θα το βάλω και σε τροπολογίες. Νομίζω ότι αφού άκουσα χθε την Επίτροπο Μάλστρομ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις ανάμεσα στις προτεραιότητε τη εμπορική πολιτική και το πώς απεικονίζεται στο προπολογισμό. Π.χ. η Κομισιόν είπε ότι θεωρούσε προτεραιότητα τη ε, μελλοντική εμπορική πολιτική, τη στρατηγική ενημέρωση ε, επικοινωνίας ε, με τους πολίτες για το τι κάνει σε εμπορικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον προπολογισμό 2005 υπήρχε μία γραμμή, ενώ τώρα ε, στον προπολογισμό του 2016 η σχετική γραμμή του προπολογισμού έχει υποστεί περικοπή. Δεν νομίζω ότι είναι συνεπέ αυτό. Δεύτερο η Κομισιόν μίλησε πολύ για, την, για το πολυμερέ επίπεδο, ότι με αυτόν τον τρόπο ασκείται η εμπορική πολιτική. Και πάλι υπάρχει μια περικοπή ε, για την πολυμερή εμπορική πολιτική. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι οι επιπρόσθετες προσπάθειες που γίνονται ε, για να υπάρξουν ε, μελέτες αντικτύπου ε, εκ των προτέρων, εκ των υστέρων και κάτι διάρκεια. Δηλαδή εξάντε εξπόστηκε να γνωρίζουμε τι, τι έχει γίνει, τι υπάρχει, να παρακολουθούμε τι γίνεται και εκ των υστέρων για να διορθώσουμε. Επίσης, θα πρέπει να επιμείνω να συμπεριλάβουμε και τις μελέτες ε, για το φύλλο. Πρέπει σε όλα όσα κάνουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, τη σημασία αυτού του θέματος. Είναι σημαντικό αυτό τον 21ο αιώνα. Επίσης, στο τέλος του 2014 είχαμε την ε, γνωμοδότηση της ΣΥΝΤΑ του David Martin και εκεί υπήρχε μία γραμμή με ένα εκατομμύριο ευρώ για να προωθήσει το δίκαιο εμπόριο. Δεν ξέρω εάν αυτή η γραμμή έχει ενταχθεί στον προπολογισμό του 2015. Θα ήθελα όμως, αν ε, υπάρχει στον προπολογισμό του 2015, να διατηρηθεί και στους ε, μελλοντικούς προϋπολογισμούς και αν όχι, να ενσωματωθεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τη συζήτηση του προπολογισμού της ΕΕ για το εμπόριο. Και ο εισηγητή ε, θίγει ένα από τα κυριότερα θέματα που και εμένα με απασχόλησαν και επικεντρώθηκα σε αυτό. Βλέποντας τις προσδοκίε ε, για την εμπορική πολιτική να μεταλλάσσονται και μια πραγματική αυθεντική ανάγκη για πληροφορίε και εμπλοκή υπάρχει ανάγκη να αυξήσουμε το δυναμικό μας και τις ικανότητές μας και αυτό είναι πρόδειλο στις συζητήσεις για την TTIP. Είναι κάτι που πρέπει ευρύτερα να εξετάσουμε. Υπέβαλα την πρόταση για πιλωτικό πρόγραμμα για να αυξηθούν τα κονδύλια ώστε να υπάρξει θετική εμπλοκή, μεγαλύτερη εμπλοκή και να είναι οι πληροφορίες διαθέσιμες να διαχέονται σε ένα ανοιχτό πλαίσιο με τον πιο θετικό τρόπο. Αυτό είναι ένα τμήμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακούγοντας τα θέματα για την πληροφόρηση υπάρχει ανάγκη να εισακούγονται οι πολίτες και τα αιτήματά τους. Όχι μόνο να διατίθενται πληροφορίες, είναι και αυτό σημαντικό. Και σε σχέση με αυτό το θέμα ένα γενικότερο ζήτημα υπαλλήλων στελέχωσης τη Γενικής Διεύθυνσης για το Εμπόριο <clears throat> και υποστηρίζουμε το αίτημα στη νέα αυτή εμπορική πολιτική που θα είναι φιλόδοξη να διασφαλιστεί αυτή η τάση. Υπάρχουν ε, αξιο, ε, υψηλού ε, επίπεδου συζητήσεις και διαβουλεύσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη και διεξάγονται και είναι θετικό το ότι βλέπουμε ο Ιγνάθιο να ασχολείται και με κάτι διαφορετικό από την TTIP αλλά δεν γνωρίζω πραγματικά τι γίνεται σε σχέση με τα στελέχη που επομίζονται όλες αυτές οι σημαντικές για μας ε, αρμοδιότητες, ε, πώς τα καταφέρνουν να είναι αποτελεσματικοί. Ίσως ε, να μπορούσαμε να το δούμε και η ίδια η Επιτροπή να προβληματιστεί για αυτό το ζήτημα πιο αποτελεσματικά και σε ένα διαφορετικό τόνο. Είναι σημαντικό νομίζω σε σχέση με προϋπολογισμό και κονδύλια η εποπτεία, η παρακολούθηση έχει ρόλο κλειδιού. Να δούμε ότι σωστά θα ε, δαπανώνται τα κεφάλαια. Έλεγχος και εποπτεία λοιπόν. Και για τη μακροοικονομική ε, συνδρομή θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους και ποιους άλλους τρόπους μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ε, ε σε τρίτες χώρες και να μην ε, υπάρχουν ε, κάποιες δυνατότητες να αναλώνονται τα κονδύλια μας ε, χωρίς να χρησιμοποιούνται για το σωστό σκοπό. Έχουμε και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ίσως οι πηχαίοι τίτλοι δεν ανταποκρίνονται στις λεπτομέρειες και σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Για μένα το εμπόριο είναι πάντα μια πολύ σημαντική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι άρρηκτα στοιχείο που εντάσσεται σε αυτή την πολιτική. Πρέπει να υπάρχει συνάφεια και συνεκτικότητα λοιπόν σε όλα, ακόμα και στο εμπόριο. Και σε σχέση και με τα δικαιώματα του ανθρώπου, στο εμπόριο επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις πτυχές και υπό το φως όλων αυτών η τελευταία παρατήρηση για την λογοδοσία σε τρίτες χώρες που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι σημαντική παρατήρηση. Δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις που να ζητούν το λόγο. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να πω στην ε, συνάδελφο την κυρία Ροντρίγκε ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Διαφωνώ που δεν υπάρχει ακόμα μία μελέτη για την επίπτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό. Επίσης, όλες οι εργασίες αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και όλες οι εργασίες της Γενική Διεύθυνση Trade να λάβουν υπόψη του τη διάσταση του φύλου. Ευχαριστώ τον συναδελφό που συνέταξε το κείμενο, τον κύριο Μπέγκε. Θέλω, να ήθελα να πω πού διαφωνούμε και πού θα παρουσιάσουμε τροπολογίες. Αυτό που στο κείμενο λέγεται φιλόδοξη εμπορική ατζέντα ή θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα φέρει ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. όπως φαίνεται από διάφορες μελέτες, θα καταστρέψει ε, θέσει απασχόληση αντί για να δημιουργήσει θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Το ίδιο και το TTIP. Ε, Επομένω, θα χρειαζόμασταν πιστώσει ε, για να κρατήσουμε αυτέ τι θέσει ε, απασχόληση λόγω αυτή τη εμπορική πολιτική που προωθείται παρά τη διαφωνία πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Ε, όταν εγκριθεί το TTIP, ε, αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη εδώ. Μπορεί επίση να έχει ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επίπτωση ε, των εμπορικών συμφωνιών στο μπάτζετ και αυτό επίσης δεν αποτυπώνεται στον προπολογισμό. Νομίζω ότι η παγκοσμιοποίηση ε, μας κάνει να χάνουμε ε, θέσεις απασχόλησης γενικά. Αυτό είναι σωστό. Η παγκοσμιοποίηση χωρίς κανόνες έφερε περισσότερη ανεργία και απώλεια θέσεων εργασιών. Επίσης, ε, όταν κανένας ζητάει οικονομική βοήθεια, χάνονται θέσεις απασχόλησης, ε, οι θέσεις απασχόλησης ε, γίνονται πολύ πιο ασταθείς κτλ. Ζητάμε επίσης περισσότερες, ε, περισσότερα χρήματα για τις αναπτυσσόμενε χώρες, περισσότερη στήριξη για, την, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα διήθησης στις τρίτες αγορές. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο David Καπλμπέρμαν που δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραβρίσκεται εδώ σήμερα το απόγευμα και μου έδωσε κάποιες ε, σημειώσει για να μεταφέρω τη θέση του σχετικά με το θέμα αυτό. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση που είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου του βεβαρημένου και ε, θεματολογίου στον τομέα του αμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ECR αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αγορές σε όλον τον κόσμο για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το ε, ε, πρότυπο κοινωνικής αγοράς που έχουμε. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει επαρκείς σπόρους ε, για να συνεχίσει όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει και άλλες μελλοντικές που μπορεί να ξεκινήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαδικασία ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ε, θα πρέπει να ζούμε εντός των δυνατοτήτων μας και να φροντίσουμε οι δημόσιοι πόροι να δαπανώνται με, ε, ανάλογα με τις αρχές αποτελεσματικότητας της λογοδοσίας και των σωστών λογαριασμών. Και γι' αυτό θα πρέπει στον προϋπολογισμό του 2016 να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή ε, αντιστοιχεία κόστους και όφελους. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, ε, το ECR έχει τρεις βασικές παρατηρήσεις. Καταρχά, το ECR δεν είναι κατά των αυξήσεων στον προϋπολογισμό για την εμπορική πολιτική. Οποιαδήποτε τέτοια αύξηση θα πρέπει να προέλθει από ανακατανομή εντός του προϋπολογισμού. Δεύτερον, όλες οι δαπάνες θα πρέπει να εξεταστούν όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και την αποδοτικότητά τους και να φροντίσουμε να δαπανώνται σύμφωνα με την αρχή της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τέλος, η μελέτη της Επιτροπής ε, για του, τους πόρους χρηματοδότησης στον τομέα του εμπορίου ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, στον τομέα αυτό είναι πολύ σημαντικό οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να ανοίξουν του λογαριασμού του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Φίλιπ Ντυποντέ από την Κομισιόν, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μπέγκε και τα μέλη της Επιτροπής σας για τις παρεμβάσεις τους και τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Γενικά νομίζω ότι οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ε, την υποστήριξη της Επιτροπής σας ε, για την εμπορική πολιτική και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις. Όσον αφορά κάποιες άλλες θα επανέλθουμε επειδή πρόκειται για πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Απαντώντας σε διάφορες θέσεις ε, που εκφράστηκαν σχετικά με την επαρκή διάθεση των πόρων, είναι σαφές ότι το όλο και αυξανόμενο θεματολόγιο στον τομέα του εμπορίου όπως το έχει παρουσιάσει ο Επίτροπος ε, αποτελεί πρόκληση. Έχει αυξηθεί πολύ και το πολιτικό ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά τα τελευταία χρόνια, κάτι που απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια επικοινωνίας και διαφάνειας από τη δική μας πλευρά. Και όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις ε, θα πρέπει να περάσουν από την κανονική νομοθετική διαδικασία και να εφαρμοστούν σωστά και να υπάρχει και σωστή παρακολούθηση για να έχουν ωφέλη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ε, ευρωπαίους πολίτες. Υπό το φως λοιπόν αυτού του φιλόδοξου θεματολογίου ε, και της κατάστασης αυτής που απαιτεί πολλούς πόρους ε, και υπό το φως τις προσπάθειες της Κομισιόν να μειώσει το προσωπικό κατά 5% κάτι στο οποίο θα συμμετέχει και η Γενική Διεθνήση Εμπορίου. Για παράδειγμα θα πρέπει να μειώσουμε κατά 21 άτομα το προσωπικό μας. Ε, εκτιμούμε την υποστήριξή σας ε, και για τους ε, πόρους εκτιμούμε πολύ την προσοχή που δίνεται όσον αφορά το δυναμικό μας και στα κεντρικά μας γραφεία αλλά και στις αντιπροσωπείες σε διάφορες χώρες. Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, όπως ανέφερα, έχει δοθεί πολύ περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό από ότι στο παρελθόν επικροτούμε το ενδιαφέρον αυτό και ήδη έχουμε αυξήσει τις προσπάθειες επικοινωνίας μας εντός των ορίων των περιορισμένων πόρων μας όπως σας ανέφερα. Για παράδειγμα έχουμε αυξήσει την διαφάνεια με την ε, δημοσίευση ε, εγγράφων, ε, είχαμε τους ε, διαλόγους με τους ενδιαφερομένους σε κάθε γύρο της TTIP. Έχουμε προσπαθήσει να αυξήσουμε την ορατότητά μας στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε περισσότερο με τους πολίτες. Επίσης είχαμε πριν τρεις εβδομάδες τις ημέρες εμπορικής πολιτικής όπου συμμετείχαν επιχειρήσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πανεπιστημιακοί. Ξέρω ότι και αρκετοί από εσά συμμετείχαν στη συζήτηση του πάνελ. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να εξηγήσουμε τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης και τη εμπορική πολιτικής μας για τους πολίτες και να απαντήσουμε σε ανησυχίες των πολιτών. Ήδη τώρα προβλέπουμε να υπάρξουν κάποιες πρόσθετες δραστηριότητε στον τομέα αυτό εντός των ορίων, εντός των περιορισμών ε, όσον αφορά το δυναμικό μας που σας ανέφερα και πολύ ευχαριστώ θα συζητήσω το θέμα αυτό μαζί σας ε, στους προσεχείς μήνες. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και το εμπόριο και την ε, συμφωνία διευκόλυνσης του εμπορίου που συνδέεται με το θέμα αυτό. Εκτιμούμε τις θέσεις σας για αυτήν τη σημαντική συμφωνία. Έχουμε διαθέσει 400 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Διευκόνησης του Εμπορίου τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2018 και μέχρι την ε, δέκατη συνάντηση και την Υπουργική Σύνοδο έχει δοθεί προτεραιότητα στη συμφωνία αυτή στα στρατηγικά έγγραφα των ε, διαφόρων ε, χρηματοδοτικών μέσων ε, και είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν επαρκή σπόροι για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Χώρες που θα χρειαστούν βοήθεια για την εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας του ΠΟΕ θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τέτοια υποστήριξη. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στη συγκεκριμένη παρατήρησή σας το Aid for Trade στον προϋπολογισμό του 2016 έχει αυξηθεί, έχει ο προϋπολογισμός ε, για αυτό και η συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού αποτελεί μικρό κομμάτι της ε, όλης προσπάθειας από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Αλλά ε, είχαμε κάποιες καθυστερήσεις λόγω κάποιων συζητήσεων που πραγματοποιούνται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιους διεθνείς οργανισμούς ε, στους οποίους συμμετέχουμε. Ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά την ε, αξιολόγηση με τους τέσσερις πυλώνες και χωρίς ε, τη συμφωνία αυτή δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση των διεθνών αυτών οργανισμών για να εφαρμόσουμε όσα είχαμε κατά νου όσον αφορά το Aid for Trade. Πολύ ευχαρίστω. Ε, θα επανέλθουμε και θα σας ε, δώσουμε γραπτές εξηγήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως άλλωστε μας ζητήσατε, με συγκεκριμένα στοιχεία μάλιστα. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις ε, σχετικά με την παγκοσμιοποίηση των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων, όπως γνωρίζετε η Κομισιόν πάντα δίνει πολύ βάρος στην κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις προσπάθειές τους να ε, εισέλθουν σε άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο και οι εμπορικές συμφωνίες δίνουν όλο και περισσότερη πρόσβαση στην αγορά για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και ο Επίτροπος ε, σας έχει διαβεβαιώσει σχετικά με αυτό. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε το ICA+, το Κόσνερ και τα ε, μέσα εταιρική σχέσης και συνεργαζόμαστε στενά με ε, οργανώσεις ε, επιχειρήσεων και τις σχετικές υπηρεσίες εντός του Κοινοβουλίου για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω, όπως είπα ήδη και πέρσι, ότι Όλα τα προγράμματα περνούν από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις με βάση τα στοιχεία. όσον αφορά την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συμμετοχή του στην εμπορική πολιτική και το θέμα της χρηματοδότησης. Όπως ε, συζητήσαμε λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και της αυξανόμενης σημασίας της εμπορικής πολιτικής. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα εμπορικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο επικροτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνομιλούμε με πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο του διαλόγου μας με την κοινωνία των πολιτών. Ενθαρρύνουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους παράγοντες να ε, εγγραφούν στο Μητρό Διαφάνειας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου και πρέπει να δίνουν στοιχεία σχετικά με την χρηματοδότησή τους. Πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμες αυτές οι πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ειδική μελέτη για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρότι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει χρήσιμες τις πληροφορίε από μια τέτοια μελέτη, ιδιαίτερα όσον αφορά τι τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, ε, που είναι αντίθετες στην εμπορική πολιτική μας. Να περάσω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα όπως είναι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και η ανάγκη για σωστή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ε, μια συμφωνίας, κάτι που συζητήσαμε μαζί σας πριν προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τα διάφορα θέματα που αναφέρονται στην ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βελτιώσει σημαντικά την αξιολόγηση και παρακολούθηση των εμπορικών συμφωνιών, ε, όπως άλλωστε τόνισε και η Επίτροπος Μάλμστρομ σε φετινή επιστολή της. Ε, θα σας κατάμε ενήμερους σχετικά με τις πρόοδου που σημειώνονται στο τομέα αυτών. Όσον αφορά την ε, πτυχή της ε, ισότητας ε, των δύο φύλων. Όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, πιστεύουμε ότι γίνονται πολλά πράγματα ήδη από το 2011 και μετά. Εξετάζεται συστηματικά η επίπτωση στην ισότητα των δύο φύλων μιας εμπορικής συμφωνίας. Και στο πλαίσιο της εισβάθος ανάλυσης εξετάζονται οι επιπτώσεις στην ισότητα των δύο φύλων και ε, στο θέμα των μη διακρίσεων στην μελέτη αντικτύπου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αυτή ακολουθείται από μία εξπόστ ανάλυση κάποια χρόνια μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου όπου συμπεριλαμβάνεται και πάλι εξέταση της ψυχής της ισότητας των δύο φύλων και επίσης ε, ε, σε όλες τις πρόσφατες εμπορικές μας συμφωνίες έχουμε κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και υπάρχουν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και εντός Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες εταίρους μας. Και επίσης, στο πλαίσιο του ε, καθεστώτος GSP, υπάρχει πρόσθετη εξέταση από πλευρά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, εξετάζουμε λοιπόν πώς μπορούν να εξαλειφθούν οι διακρίσεις εις βάρος γυναικών και εξετάζουμε τα στοιχεία που παρέχονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να εξηγήσετε σα παρακαλώ περισσότερο το θέμα Aid for Trade, την ε, βοήθεια ε, και σε σχέση με τι εμπορικέ συμφωνίε. διότι δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Ναι. Για την ε, γραμμή του προπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου για το Aid for Trade, πολύ, πολύ πολλή από αυτή τη βοήθεια πηγαίνει σε διεθνείς οργανώσεις. Δίνουμε κονδύλια σε διεθνείς οργανώσεις και μαζί τους ε, υποστηρίζουμε κάποιες χώρες ε, που το έχουν ανάγκη μέσω αυτής της γραμμής προϋπολογισμού. Με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού η Κομισιόν ζήτησε αυτές οι οργανώσεις να δώσουν κάποια στοιχεία στο ό,τι αφορά την αξιολόγηση των τεσσάρων πυλών για να δείξουν ότι μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα κονδύλια στο εσωτερικό τους, να σεβαστούν κάποιες βασικές γραμμές που αναφέρει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Κάποιες από αυτές τις ε, διεθνείς οργανώσεις ε, έχουν συζητήσει μαζί μας, αλλά οι συζητήσεις αυτές ε, καθυστέρησαν, ήταν δύσκολες, ειδικά με τον Οσάφερ Φερρυπίν. Και μόνο πρόσφατα ε, μπορούμε να πούμε ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αλλά δεν σημειώθηκε αρκετά έγκαιρα όταν προετοιμαζόταν ο προϋπολογισμός. Και μάλιστα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Η Γενική Διεύθυνση ε, Προϋπολογισμού και η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ε, ολοκληρώνονται, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές τι συζητήσεις πριν βάλουμε τίποτα εμείς στον ε, επιχειρησιακό μας προϋπολογισμό, στο δικό μας προϋπολογισμό. Μάλιστα. Όλα αυτά που συζητάμε, ε, το γεγονός ότι συζητάμε διμερείς εμπορικές συμφωνίες, μπορεί να είναι πρόβλημα για το κοινό. Ε, εάν δεν είναι προς, το όφελος των, ε, λιγότερων επιτυγμένων χωρών και ταυτόχρονα μειώνουμε ε, τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα για το εμπόριο. Θέλετε το λόγο. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω. Ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, <clears throat> μας διασφάλισε ότι θα δοθούν αποσαφηνήσει αυτήν την εβδομάδα. Ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι τα προηγούμενα έτη υπήρξε πρόβλημα. Αφενός, <clears throat> σε πολλούς τομείς, διεθνώ είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός και στι δραστηριότητε των Ηνωμένων Εθνών και ως αρχή επί του προπολογισμού, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, <clears throat> συχνά ποτέ δεν, επαρ... δεν ενημερωνόμεθα επαρκώς. Κατ' το παρελθόν δεν είχαμε πρόσβαση στα audits, στους ελέγχους δηλαδή των ε, Ηνωμένων Εθνών, ενώ τα κράτη-μέλη είχαν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και στοιχεία και γνωρίζουμε ότι δεν πήγαν όλα 100% όπως τα θέλαμε. <clears throat> Κατανοούμε πολύ καλά την προσεκτική και συνετή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα προσέξει να δει αν εκείνοι που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση αυτών των θεμάτων Στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρούν τους κανόνες και κανονισμούς μας. Πρέπει να δούμε όμως και ελπίζω ότι θα υπάρξουν περαιτέρω πληροφορίες που θα μας δώσουν αυτή την εικόνα αν <clears throat> ενδεχόμενα συμπληρωματικά κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν ώστε και πάλι να μπορέσουμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν δυνατότητες τι συμβαίνει ακριβώς και να μπορούμε έτσι με ήσυχη συνείδηση να δώσουμε το πράσινο φως για να προχωρήσουν αυτά. Αυτό είναι μία από τι δυνατότητε που πρέπει να επιφυλαχθούμε αυτών ώστε να δοθεί ένα πολιτικό μήνυμα. Ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει και να έρθουμε στο ύψο των υποχρεώσεών μα, αλλά σύμφωνα με τι πληροφορίε που πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μα, να δούμε τι γίνεται. Σε σχέση για παράδειγμα με τον ΩΣΑ. αν υπάρχουν εδώ προβλήματα ή κάποιε δυσκολίε να δοθεί το καλό παράδειγμα, αλλά τουλάχιστον να δούμε του κανονισμού και διατάξει. Δεν είναι δυνατόν αφενό ε, να ζητούνται κονδύλια και κατά το τέλη του έτους ε, εμείς ως αρχή του προϋπολογισμού να πρέπει να ε, συνενέσουμε σε κάτι για το οποίο μπορεί ίσως να μην έχουμε ενημερωθεί επαρκώς. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Προθεσμία 17 Ιουλίου για τις τροπολογίες. Και για τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό 3 Αυγούστου. 31 Αυγούστου θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές. Πολύ καλά λοιπόν. Και στη συνέχεια ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο, το σημείο 18 της ημερήσια διάταξης. Εχθές και σήμερα είχαμε αρκετές φορές το θέμα του ΠΟΕ και των εξελίξεων σε σχέση με τον ΠΟΕ. Γνωρίζουμε σε σχέση με τη διάσκεψη του Μπάλι ήταν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, τι απέρευσε και γνωρίζουμε επίσης ότι μέχρι σήμερα μια νέα εντολή ζητείται για τη διάσκεψη στην Κένια κατά τον μήνα Δεκέμβριο που δεν έχει ακόμα τεθεί επί τραπέζης ε, ώστε να ε, λειτουργήσει όπως πρέπει και γι' αυτό έχει νόημα και είναι αναγκαίο κάπως να μπορέσουμε να ασκήσουμε πιέσεις για να προαθεί αυτό και να υπάρξει μια σαφή τοπο, τοποθέτηση για την ε, δική μας ε, κοινοβουλευτική παρουσίαση των θεμάτων. Τι επιθυμούμε εμείς δηλαδή να γίνει σε σχέση με αυτή την υπουργική διάσκεψη στην Κένια το Δεκέμβριο όπου θα εκπροσωπηθούμε και εμείς σε αυτήν. Κατά τούτο λοιπόν θα ρωτούσα τους συναδέλφους τώρα. Έχουν συγκεκριμένες προτάσεις να καταθέσουν για το ψήφισμα. Για αυτό το ψήφισμα θα συζητήσουμε στις 22 Σεπτεμβρίου και θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως όμως από δική σας πλευράς, με βάση τη συζήτηση εχθές και σήμερα, υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις που θέλετε να καταθέσετε. Κύριε Μπούχνερ, εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή και που μου δίνετε τον λόγο τώρα. Θέλω κάποια σύντομη, πολύ σύντομη παρατήρηση να κάνω. Είναι σημαντικός ο γύρος της Δόχα να είναι ένας αναπτυξιακός γύρος διαβουλεύσεων. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο αυτών των διαπραγματεύσεων. Μέχρι στιγμής ε, δεν ήταν αυτό κάτι πρόδειλο και δεν γινόταν έτσι αυτόματα συχνά συμβαίνει η επιθυμία των ιδιωτικών επιχειρήσεων να, να έχει τύχη να βρίσκονται στο προσκήνιο. Η ημερήσια διάταξη σε σχέση με θέματα όπως τρόφιμα και ασφάλεια τροφίμων και επισητιστικής ε, ασφάλειας θα πρέπει να δούμε τα θέματα των γεωργικών αυτών προϊόντων και τροφίμων που έχουν πολύ ε, έντονη επιδότηση και υποστηρίζονται χρηματοοικονομικά στην Ευρώπη εις βάρος των αναπτυσσομένων χωρών. Πρέπει να καταστεί σαφές γιατί σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν ακριβώς πολύ μεγάλες επιφυλάξει για αυτή την κατάσταση. Καλό θα ήταν λοιπόν να, δίναμε, να προωθούσαμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κέντρο βάρους ε, σε σχέση με την ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές πτυχές. Άλλα θέματα σε σχέση με το ψήφισμα αυτό που θα θέλατε να εντάξουμε. Δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις. Θα δώσω τον λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παύλο Γκρατσότη παρακαλώ. Thank you, um, in the in Η κατάσταση στη Γενέβη όπως ε, ίσως μάθατε από τον τύπο ή ακούσατε χθες, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Υπάρχουν ε, δυσκολίες από πλευράς να συμφωνήσει με το πρόγραμμα εργασίας που προτείνει το Γενικό Συμβούλιο για να εγκριθεί μέχρι τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει συμφωνία λοιπόν επένδυνος εγγράφου, αλλά αυτό δεν μας ε, αποτρέπει από το στόχο μας που είναι να βρούμε μια τελική συμφωνία στο Ναϊρόμπι στο τέλος του 2015. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση ενώ υπάρχει διαφωνία. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και μια ισορροπία που θα απεικονίζει τη σημερινή κατάσταση και κυρίως τις διστάμενες απόψεις των μελών του ΠΟΕ, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών, των αδειωμένων οικονομιών και των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Είναι η πρώτη Υπουργική Σύνοδος που γίνεται στην Αφρικανική Ήπειρο, η Ήπειρος η οποία έχει και τις περισσότερες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια σημασία σε αυτές τις χώρες. Περιμένουμε τις ιδέες σας και μια πολιτική καθοδήγηση από σας. και το πού θα σταθούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ο στόχος είναι να ολοκληρώσουμε πολιτικά το DDA, το γύρο της τη συμφωνία της Ντόχα. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί ο ΠΟΕ να χάσει τη σημασία του και να χάσει τον κεντρικό ρόλο που θα πρέπει να έχει και ως βασικού εγγυητή για αυτές τις μικρές και ευάλωτες οικονομίες που δεν έχουν τα μέσα και τις διασυνδέσεις να, να διαπραγματευτούν μεγάλες ε, διμερείς και πολυμερείς ε, συμφωνίες. Αυτό θα χρειαστεί, θα απαιτήσει δέσμευση από μεγάλους εταίρους, με μεγάλους παίκτες, εμείς είμαστε ένας από αυτούς, αλλά και άλλες δύο οικονομίες θα πρέπει να συνεισφέρουν. Περιμένουμε λοιπόν την ε, καθοδήγησή σας και ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε βασικό, θεμελιακό το ερώτημα. Στη Γενέβη υπήρχε μια αισιόδοξη άποψη, αυτή το Φεβρουάριο ακούστηκε, ότι τον Ιούλιο θα υπήρχε το κείμενο για μια αναθεωρημένη διαπραγματευτική εντολή. Αυτό θα είναι σημαντικό για την Υπουργική Συνάντηση της Κέννη. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει εντολή όμως. Δεν υπάρχει κείμενο. Ποια είναι η αποψή σα στην Κομισιόν, πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ρεαλιστικός πόσο η δυνατότητα να ετοιμαστεί κάτι, ένα κείμενο, πριν ξεκινήσει η σύνοδος της Κένια. Ευχαριστώ. Υπάρχει η δυνατότητα φυσικά. Αυτό που λείπει τους τελευταίους 6 μήνες είναι μια σαφής κατανόηση από όλα τα μέλη ότι η συμφωνία που μπορούμε να πετύχουμε στο Ναϊρόμπι σε καμία περίπτωση δεν είναι μια συμφωνία όπως αυτή που είχαμε φανταστεί το 2008 της, ε, την τελευταία φορά που είχαμε διαπραγματευτικά κείμενα στο τραπέζι. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό πια. Γιατί άλλαξε η διαπραγματευτική κατάσταση. Και γιατί άλλαξε η παγκόσμια οικονομική ισορροπία. Και για το πώς ε, λειτουργεί το παγκόσμιο εμπόριο. Εάν αυτή η αλλαγή δεν καταγραφεί στα μυαλά όλων, δεν θα έχουμε συμφωνία. Εμείς προσπαθούμε να το πετύχουμε αυτό. Είχαμε πει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο προς τη σημερινή πραγματικότητα. Και ίσως να, μειώσουμε, να χρειαστεί να μειώσουμε και το βαθμό φιλοδοξίας μας. Ε, και το επίπεδο απελευθέρωσης που θέλαμε στο παρελθόν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κράτη τα οποία είναι προσκολλημένα στο κείμενο με βάση το οποίο διαπραγματευόμαστε το 2008. Οι πιο προσκολλημένοι, παραδόξως, είναι αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την αποτυχία των διαπραγματεύσεων τότε και απέρριψαν το κείμενο το 2008 και απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις. Παράδοξα, αλλά συμβαίνουν αυτά. Χρειαζόμαστε μια γρήγορη κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Εάν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, όπως είπα, κινδυνεύουμε να μην υπάρξει μια πολιτική ε, συμφωνία για το γύρο της Δόχα. Το, το Σεπτέμβριο οι αντιπροσωπείες θα προσπαθήσουν να βρουν σε περίπτωση που δεν υπάρξει παγκόσμια συμφωνία, μια κάποια συμφωνία. Αλλά αυτό θα κοστίσει και, στη, και στην οργάνωση και, στην, και στον κύριο της Δόχας. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Αλλά μπορώ να πω και σε άλλες λεπτομέρειες, αν το επιθυμείτε. To, be honest, To be honest, I'm not that is. Ειλικρινά, δεν είμαι πολύ βέβαιος σχετικά με αυτό, Χέλμουτ. Και εγώ θα ήθελα να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Να ξαναρωτήσω λοιπόν, υπάρχει η δραματική έκκληση του Γενικού Διευθυντή του ΠΟΕ που έκανε τον Ιούνιο, που κάλεσε όλα τα κράτη να σκεφτούν προς ποια κατεύθυνση κινούνται. Και θα με ενδιέφερε σε πείσμα όλων των ε, διαβεβαιώσεων ε, της ε, κυρίας Μάλμστρομ να γνωρίζω, υπάρχει κοινή προσέγγιση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουμε. Εδώ και δέκα χρόνια ή ακόμα περισσότερο ε, διαπραγματευόμαστε. Γνωρίζουμε λοιπόν προς τα που κινούνται τα πράγματα. Πού βρίσκονται οι πραγματικές δυσκολίες. Πού θα πρέπει να πετύχουμε συμβιβασμούς. Η ουσία πού βρίσκεται. Και θα ήθελα να προσθέσω την ερώτηση ποιες χώρες είναι ιδιαίτερα προβληματικές και ποιε προορατικέ. Είχαμε την εντύπωση το Φεβρουάριο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη συνεργάζονται πολύ στενά μεταξύ τους. Αυτό συνεχίζει να ισχύει. Και ποιος εμποδίζει την πρόοδο. Και η Έμα έχει μια ερώτηση ακόμα. Ναι, νομίζω ότι πολλοί είμαστε δυσαρεστημένοι που δεν υπάρχει ε, συμφωνία και κίνηση από πλευράς ε, των μελών ε, του ΠΟΕ. Θα ήθελα να είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο κοντά σε μια συμφωνία κατά την Υπουργική Διάσκεψη, αλλά ιδιαίτερα στο Ναϊρόμπι. Δεν θα ήθελα πάρα πολύ να δω να κάνουμε σόου στην Κένια, αλλά με πολύ ισχνό αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου χρήσιμο. Μήπως μπορείτε λοιπόν να σχολιάσετε, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να ενθαρρύνουμε τους άλλους να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να πάμε στην Κένια γνωρίζοντας ότι, κάταμε, ότι κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής το βασικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι αυτό που συνδέεται με τους εγχώριους παραγωγούς στη Γεωργία. Αυτό, καλός ή κακός, είναι κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πολλά, διότι έχουμε ήδη κάνει πάρα, ε, έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά. Έχουμε ε, αναμορφώσει την ε, γεωργία μας, έχουμε μειώσει τις ε, ενισχύσεις. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Είμαστε ο καλός μαθητής, στον οποίο όμως δεν δίνει πολύ προσοχή ο δάσκαλος. Ε, άλλες ε, χώρες δεν κάνουν εξίσου πολλά. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα νομοσχέδιο για τη γεωργία, το οποίο σύμφωνα με αρκετές μελέτες δεν θα τους επιτρέψει να δεχτούν το κείμενο του 2008. Και ακόμα χειρότερα η Κίνα στρεβλώνει τις ενισχύσεις, ενώ ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει μόνο ένα όριο de minimis. Δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα να ταπανίσει όσα η Βραζιλία ή η Ινδία, γι' αυτό δεν κάνουν πολλά. Γι' αυτό, όπως έχει εξηγήσει ένα αυστραλέζο καναδικό κείμενο, παρότι πολλοί δεν ε, προσφέρουν ενισχύσει άνω του 20-25% του ορίου δηλαδή, πολιτικά βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δεν ε, θέλουν να στελέψουν τα περιθώρια τους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν απόλυτα σαφείς ή ε, ούτε η Κίνα πρόκειται να μετακινηθεί και η Κίνα θεωρεί απαράδεκτα τα αιτήματα στον τομέα αυτόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει λύσεις που να μπορεί να προβάλλει για να σημειωθεί πρόοδος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο πρόβλημα συνδέεται με την πρόσβαση στις αγορές. Και εδώ έχουμε μια διπλή δυσκολία από τη μία, πολλοί παράγοντες εντός του ΠΟΕ ε, ε, διμερώς και περιφερειακά ε, έχουν απελευθερώσει σε σημαντικό βαθμό το εμπόριο και γι' αυτό δεν θέλουν απελευθέρωση σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε τον παράγοντα Κίνα, διότι απελευθέρωση σημαίνει άνοιγμα σε προϊόντα από την χώρα που παράγει το 50% των μεταποιημένων προϊόντων του κόσμου. Αυτές λοιπόν είναι δυσκολίες δεν αποτελεί εμπόδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε προτείνοντας κάτι ε, αξιόπιστο το οποίο να ταιριάξει με τις επιθυμίες όλων. Σαφές είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η έλλειψη πολιτικής βούλησης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πετύχει ακόμα το στόχο μας. Το χρονοδιάγραμμά μας δείχνει ότι απομένουν ακόμα πράγματα να γίνουν. Είχαμε ένα σημαντικό πολιτικό ραντεβού διατλαντικό και ελπίζουμε το Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να ασκήσουμε ισχυρή πίεση ώστε οι πρωτεύουσες ή οι υπουργοί να πετύχουν σημαντικό αποτέλεσμα στο Ναϊρόμπι. Είναι πρώτη φορά που πάμε στην Αφρική και θα είναι κρίμα εάν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία. Πρόκειται για πολυμερείς διαπραγματεύσεις με πολλούς παράγοντες και δυστυχώς υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει την επίτευξη καλού αποτελέσματος. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν, ε. Ωραία. Κλείνω λοιπόν το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Και προχωράμε τώρα στο σημείο 19. Εδώ μας ενδιαφέρει η εξοδαφική νομοθεσία. Πρόκειται για αναδιατύπωση. Ο David Μάρτιν είναι εισηγητής μας και του δίνω το λόγο. Thank you. As you say, this is the... Ευχαριστώ. Πρόκειται για την αναδιατύπωση όσον αφορά την εξοδαφική εφαρμογή νομοθεσίας πρόκειται για τέτοια θέματα όπως κυρώσει τον ΗΠΑ για παράδειγμα όσον αφορά στην Κούβα, Λιβύη και άλλες χώρες που επιβάλλονται σε άτομα και που ε, έχουν επιπτώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τις εξοδαφικές αυτές πράξεις θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και έτσι λοιπόν το 1996 όταν είχαμε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και για την προστασία <clears throat> ε, ε, επιχειρήσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα έπρεπε να υφίστανται τέτοιου είδους ε, καθεστώτα καθώς επίσης και το τι θα γινόταν σε σχέση με Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τέτοιου είδους διατάξεις ήταν επιζήμιες για αυτούς σε σχέση με τις ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις ε, και τις, την μη αλλίωση των πλαισίων αυτών πρόκειται για μια πολύ θετική συγκυρία για τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων γιατί είχαμε τις κινήσεις για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ ΙΠΑ και Κούβας και σήμερα το πρωί φυσικά και τη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Υπηρεσία Εξωτερικής, Εξωτερικών Δράσεων αν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σχετικά και να δούμε πώς είναι δυνατόν αυτού του είδους ε, τα θέματα να μειωθούν σε εμβέλεια τα επόμενα χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ρώτησα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπήρχαν κάποια προβλήματα σε σχέση με τις διατάξεις της TTIP και τι θα σήμαινε η εξοεδαφική εφαρμογή τέτοιων διατάξεων σε σχέση με επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούγαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις TTIP τι ε, συμβαίνει ακριβώς. Ακούμε καμιά φορά φήμες ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όπως η Αυστριακή για παράδειγμα τράπεζα, η AG τηλεφωνικά που έλαβαν απαιτήσει από πλευρά της, ε, τον είπα να σταματήσουν ε, την εμπλοκή τους και τις ε, σχέσεις τους με την Κούβα. Σε σχέση με την ισχύ τέτοιων διατάξεων θεωρούμε ότι δεν υφίσταται και ότι είναι άκυρες. Πρόκειται λοιπόν για μια αναδιατύπωση ουσιαστικά και θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο θα έπρεπε να είναι προσπελάσιμο σε σχέση με τα άτομα, να είναι άτομα, να είναι κατανοητό και εύληπτο. Και ε, υπήρξε εργασία ακριβώ για αυτή την αδιατύπωση ώστε να υπάρξει βελτίωση του κειμένου, να είναι πιο εύληπτο. Ποια είναι τα θέματα. Πρώτα, το μεγαλύτερο θέμα για μένα είναι η νομική βάση. Χρησιμοποιούνται τρεις νομικές βάσεις. Το 207 για την κοινή εμπορική πολιτική και το άρθρο 64 για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Και είναι απόλυτα ε, λογικά τα πλαίσια αυτά. Επίσης ζητείτε να υπάρχει η ρήτρα ευελιξίας, ε, το 352 δηλαδή άρθρο. Και εδώ δημιουργούνται ίσως ε, κάποια, κάποιες ανησυχίες είναι αναγκαίο για παράδειγμα να συμβαίνει αυτό μια και τα άλλα άθρα επαρκούν πλήρως και θεωρεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι η επάρκεια αυτή είναι δεδομένη. Καλό είναι να μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί το 352 άρθρο και νομίζω ότι και εσωτερικά αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί αναφέρθηκε από κυβερνητικέ πηγές ότι οτιδήποτε απαιτεί ε, πρωτογενή νομοθεσία και το 352 θα απαιτούσε κάτι ακόμα και αν πρόκειται μόνο για θέμα αναδιατύπωσης οποιαδήποτε αλλαγή αυτής ε, της φύσης σε σχέση με το 352 θα απαιτούσε πρωτογενή ε, νομοθετική ρύθμιση από πλευράς ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Και υπάρχει λοιπόν εδώ και ο κίνδυνος της χρήσης του 352 αν συνεπάγεται τέτοιες συνέπειες. Και πρέπει να δούμε γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πρόκειται για μια τεχνική αλλαγή και εισάγονται οι κατεξουσιοδότηση πράξης όσον αφορά τις κυρώσεις και πάλι εδώ θα ήθελα να μας επεξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι αυτά τα κριτήρια των κατεξουσιοδότηση πράξεων εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με την εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου υπό το άρθρο 7 του κανονισμού απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει άμεσα και πλήρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κυρώσει τρίτων χωρών ει βάρο των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πότε συνέβη κάτι τέτοιο για τελευταία φορά. σω θα έπρεπε να το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδιαφέρον θα ήταν να ακούσουμε το τι συμβαίνει. Και χρήσιμο θα ήταν θα, αν θα μπορούσε να συνοψίσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τα συμπεράσματα των πιο πρόσφατων ε, ερευνών που έγιναν και πότε θα αναμέναμε μια νέα έκθεση το δυνατόν ταχύτερα γιατί πρόκειται για ένα ε, θέμα το οποίο είναι περίπλοκο αλλά θα μπορούσε να ε, μπορέσει να ρυθμιστεί και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ David Martin. Ο μόνος κοιόδης εισηγητής παρόν είναι ο κύριος Μπούχνερ. Θα ήθελε να παρέμβει. Δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω. Όπως ε, ακριβώς προηγούμενα αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα νομικά θέματα δεν νομίζω ότι στο, στον πολιτικό τομέα, στο πολιτικό επίπεδο μπορούν αυτά να επιληθούν. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν πιο εξειδικευμένα να διευθετηθούν αυτά. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα λάβει τον λόγο. και εσείς μετά στη συνέχεια. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman. Um, I see several different questions. Βλέπω ότι υπάρχουν διαφορά, διαφορετικά θέματα εδώ που εντάσσονται. Και εγώ ως μέλος της, ε, των νομικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και υπεύθυνο για την, τα θέματα διατύπωσης θα έπρεπε να τοποθετηθώ σε κάποια από αυτά τα θέματα, εκείνα που αφορούν τα νομικά ζητήματα φυσικά και ιδιαίτερα σε εκείνο το θέμα που αφορά την νομική βάση ακριβώς αυτής της πρότασης, αυτής της πράξης και την επιλογή των κατεξουσιοδότηση πράξεων για την εισαγωγή των αναγκαίων αλλαγών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ με κάθε συντομία στους λόγους για τους οποίους εμείς προτείνουμε αυτή την αναδιατύπωση, αυτή την πράξη. Πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικού χαρακτήρα εγχείρημα μέσα στο πλαίσιο του Trade Omnibus όπως το αποκαλούμε. Τι είναι το Trade Omnibus. Πρόκειται για δύο κανονισμούς. Τον κανονισμό 37 και τον κανονισμό 38 του 2013 και μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ως παράτημα προσαρτηθεί σε αυτούς τους κανονισμούς. Θα έπρεπε πιθανότατα να σας αναφέρω από αυτό το κείμενο τα σε σχέση με το 2013 η υιοθέτηση αυτού του κανονισμού θα συνεπάγεται σημαντικό αριθμό τροπολογιών, τροποποιήσεων στις νομικές πράξεις για να βελτιωθεί λοιπόν το κείμενο αυτών των πράξεων θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κωδικοποίηση αυτών των νομικών κειμένων. Μόλις θα, έχει, θα εγκριθεί αυτός ο κανονισμός, δηλαδή ο 37 του ε, αντίστοιχου έτους. Λοιπόν, βασικά τι κάνουμε. Ξεκινήσαμε την κωδικοποίηση αυτή το 2.21 του 1996 αλλά αμέσω κατέστη σαφές ότι κάποιες ε, μικρές αλλαγές θα έπρεπε να εισαχθούν και να γίνουν όσον αφορά το άρθρο 5 αυτού του κανονισμού. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να μετατρέψουμε την κωδικοποίησή μας σε μια αναδιατύπωση. Και αυτό επισημάνθηκε στο σημείο 4, στο εδάφιο 4 του επεξηγηματικού μνημονίου Explanatory Memorandum. Λοιπόν, τώρα, των λεχθέντων. Σύντομα θα ήθελα να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις που διατυπώθηκαν για τα κυριότερα νομικά ζητήματα που αφορούν αυτή την πρόταση αναδιατύπωσης. Καθώς αφορά τα ίδια η νομική βάση, η απάντηση είναι σχετικά απλή. Όπως προανέφερα, πρόκειται για ένα, μια άσκηση κωδικοποίησης, ένα εγχείρημα πρωτοβουλία κωδικοποίησης που μετατράπηκε σε μια αναδιατύπωση για καθαρά τεχνικούς λόγους. Αλλά όπως κατέστησε συνέχεια σαφέσα από την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση του Trade Omnibus, <clears throat> έπρεπε όλες οι νομικές πράξεις να κωδικοποιηθούν όσες καλυπτόντουσαν από το Trade, trade Omnibus. Γι' αυτό θα μπορούσαν όλα αυτά να εξεταστούν μέσα σε ένα πλαίσιο κωδικοποίησης. Και αυτό το οποίο είναι θεμελιώδες και πρέπει να υπογραμμιστεί όσον αφορά κωδικοποίησης, τι είναι. Είναι το ότι υπό τις ε, ε, εφαρμοστές διατάξεις σε σχέση με τη διοργανική συμφωνία δεν μπορούν να εισαχθούν κάποιες θεμελιώδεις ουσιώδεις αλλαγές σε ένα νομικό κείμενο το οποίο ε, κωδικοποιείται. Και έτσι λοιπόν εφαρμόζοντας αυτή την αρχή θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να διατηρήσουμε την ενισχύ αρχική νομική βάση που αναφερόταν στο άρθρο, στον κανονισμό 221 του 1996. Ε, Τότε, εκείνη τη χρονική στιγμή, τα άρθρα του κανονισμού που χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για την έγκριση, χρησιμοποιήθηκαν ως νομική βάση για την έγκριση αυτής της νομικής πράξης. 73 γ, εδάφιο γ, 113 και 235 της συνθήκης της ε, δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ίσας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μια και θεωρήθηκε ότι αυτά τα άθρα ήταν η νομική βάση για τον ενισχύ κανονισμό, έπρεπε στη συνέχεια απλά να αναπαράξουμε αυτά τα άθρα στην ε, πράξη αυτή, μετατρέποντάς τα τα άρθρα τα οποία ε, είναι τα εφαρμοστέα άρθρα αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση. Αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο τρία διαφορετικά άρθρα της συνθήκης προτείνονται ως νομική βάση για, αυτή την, το, για αυτό το εγχείρημα αναδιατύπωσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί όλα αυτά και τα τρία άρθρα να χρησιμοποιούνται ως νομική βάση και τα τρία. Το αντίθετο, οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από με τις νομικές υπηρεσίες και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με προσοχή εξετάζουν τώρα τη νομοδότηση που συντάχθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κοινοβουλευτική Επιτροπή, για την ενδεδειγμένη νομική βάση που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και μπορώ να θεωρήσω ότι και οι τρεις ε, νομικές υπηρεσίες επί της αρχής συμφωνούν σε σχέση με τη γνωμοδότηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Και έτσι ομολογούμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο η νομική βάση η οποία τελικά θα μπορούσε να επιλεγεί θα μπορούσε και να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας. Και μετά όσον αφορά τις αλλαγές, την αλλαγή που προτείνεται σε σχέση με το άρθρο 5. Όπως προανέφερα, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αυτό το εγχείρημα μετατράπηκε από μια κωδικοποίηση σε μια αναδιατύπωση. Εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε τελικά καθοριστικά την εντύπωση ότι η λησβονοποίηση των ενισχύ κανόνων μέσω του εγχειρήματο Trade Omnibus δεν ήταν κάτι πλήρες ε, ως εγχείρημα. Κάτι είχε αμεληθεί σε σχέση με το άρθρο 5 για παράδειγμα. Και από τις αναφορές ε, που ε, συμπεριλαμβανόντουσαν στα άρθρα 5, 7 και 8 μπορεί κανείς εύκολα να συναγάγει ότι υπήρχε μία πρόθεση να χρησιμοποιηθούν κατά εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά την αδειοδότηση που θα δινόταν σε άτομα για να μπορέσουν να ε, συμμορφωθούν και ευθυγραμμιστούν με αυτές τις απαιτήσεις... Ε, καθώς είναι σαφές από τα ε, κείμενα που εγκρίθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 8, καθώς επίσης και τις αναφορές που εμπεριέχονται στο άρθρο 7. Όμως ποια είναι η ουσία εδώ το κύριο ζήτημα. Είναι ότι είχαμε την εντύπωση ότι το ζήτημα πώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί η θέσπιση κριτηρίων που θα ίσιαν όσον αφορά αυτές τις εξουσιοδοτήσεις δεν είχε επαρκώς ρυθμιστεί, δεν είχε επαρκώς καλυφθεί. Ιδιαίτερα κατά την χρονική στιγμή της εγκρίσεως της ε, πρωτοβουλίας Trade Omnibus. Η πρώτη μας αντίδραση λαμβάνοντας υπόψη αυτό ήταν η εφαρμογή της γενικής, των γενικών αρχών που απορρέουν σε σχέση με την Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό και τα όρια των εφαρμοστέων εφαρμοστικών πράξεων και των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Και υπό τις τρέχουσες διαδικασίες ε, θεωρείται ότι όταν πρόκειται για την θέσπιση κριτηρίων αυτό θεωρείται ως διεργασία ως κάτι το οποίο συνιστά μια συμπληρωματική δραστηριότητα. Δραστηριότητα που συμπληρώνει το ενισχύει υφιστάμενο νομικό κείμενο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει αυτό να γίνει μέσω κατεξουσιοδότησης υπάρξεων. Ίσως απλά θα έπρεπε εδώ να σας αναφέρω και κάτι άλλο, το ότι αυτή η πρακτική είναι κάτι το οποίο αναφέρεται επίσης και σε ένα πολύ πρόσφατο κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο, μια πρόταση για την κοινή προσέγγιση των κατεξουσιοδότηση πράξεων, που ως παράδειγμα της νέας διοργανικής συμφωνίας για, την για το καλύτερο νομοθετικό έργο έχει προβλεφθεί. Το σημείο 8 αυτής της κοινή προσέγγισης ερμηνείας ή κατανόησης αναφέρει ότι σε παρόμοιες καταστάσεις η επιλογή μας θα ήταν η πρόταση κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Ευχαριστώ. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν αυτή τη σαφή εξήγηση. Για τα πολιτικά θέματα, ποιο θα μα μιλήσει, ο Ντέιβιτ. Καλή η απάντηση τη Κομισιόν, αν κατάλαβα καλά. Συμφωνούμε για την αλλαγή της νομικής βάσης ή για τακτικούς λόγους η Κομισιόν ε, πρότεινε τρει νομικέ βάσει, αλλά δεν έχει πρόβλημα με τη διαγραφή του 352. Τη νομική βάση 352. Για τι κατεξιοδότησει πράξη Κατεξιοδότηση πράξη. Άκουσα την, εξέ, την εξήγηση τη Κομισιόν. Εμεί από πλευρά Κοινοβουλίου δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα κάνει το Συμβούλιο βέβαια αν θα τη δεχτεί. Οπότε εγώ είμαι εντάξει με τις εξηγήσει. Ωραία. Περιμένω το σχέδιο εκθεσής σας στις 19 Νοεμβρίου. Τροπολογίες ε, για τις τροπολογίες έχουμε προθεσμία μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Επόμενο σημείο είναι το σημείο 20. Εκθέσεις παρακολούθησης ή μάλλον εκθέσει των ομάδων παρακολούθηση, διορθώνει ο πρόεδρο. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο κανονικά για κάτι τέτοιο, αλλά θα ζητήσω. Να ακούσετε, να ακούσετε τα σχόλιά σας. Δεκατασιωτέος γύρος για το Τίζα. Για το Μερκοσούρ και Σάλβα, έχετε να μας πείτε κάτι. Πάμπλο. Για το Μερκοσούρ. Τι έχει να πει η ομάδα παρακολούθηση. Ναι, στι 23 Ιουνίου κάναμε μια συνεδρίαση με τον Ματία Γιούργκεσεν. Σας είχα πει όλα αυτά που ξέραμε ότι κατά την Υπουργική συνεδρίαση η ε, συνεδρίαση η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Υπουργούς του Μεξικού και με τη ΣΕΡΛΑΚ υπουργοί αποφάσισαν για το πώς θα εξασφαλίσουν την αλλαγή, πώς θα προχωρήσουμε την ανταλλαγή διαπραγματευτικών θέσεων. Υπάρχει συνεχής επαφή με τις εθνικές αρχές. Από τη Βραζιλία πήγε στην Παραγουάη η Προεδρία τον Ιούλιο και ο Ταβάρε Μπάσκες ο Κορτές έχουν υποβάλει ε, χρονοδιάγραμμα για να σταματήσουν οι μη δασμολογικές, τα μη δασμολογικά εμπόδια που προ... το διασυνοριακό εμπόριο. Η Παραγουάη, συγγνώμη, η Αργεντινή ζητάει περισσότερο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Η Βενεζουέλα αποφάσισε να μην πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία και η Βολιβία απορρίπτει τη θέση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ και απειλεί ότι αν υπογραφεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου δεν θα, θα φύγει από το Μερκοσούρ η Βραζιλία και η Παραγουάη θα πρέπει να υπογράψει ούτως ώστε η Βολιβία να γίνει το έκτο μέλος του Μερκοσούρ. Τα επόμενα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τι διαπραγματεύσει με βάση την παλιά εντολή. Είπε όμως ότι δεν θα δημοσιευτεί αυτή. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να, να προβούν σε ανταλλαγές ε, προσφορών, ε, πρόσβαση στην αγορά, ε, ίδια επίπεδα φιλοδοξίας, και να υπάρξει μια ανταλλαγή θέσεων προσφορών μέχρι το τέλος του 2015. Οι αγιοργικές πολιτικές είναι προφανώς το βασικό εμπόδιο. Και η Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτιάξει ένα κατάλογο με αγαθά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η Παραγουάη θα μπορούσε να δώσει μια όθηση σημαντική, ούτως ώστε να υπογραφεί η συμφωνία μέσα στο 2016. Αυτή είναι η κατάσταση και αν έχετε ερωτήσεις εδώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην Ρωσία-Ουκρανία, κύριε Λαντσπέρκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι είχαμε συνάντηση της ομάδας παρατηρητών μαζί με ε, το, τους ε, Φινλανδούς συναδέλφους μας ε, για την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η βασική συζήτηση έγινε για την τριμερή συνάντηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία και Ουκρανία. Τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ε, συζήτησης πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών, διότι οι διαπραγματεύσεις ε, συνεχίζονται. Γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Τα βασικά θέματα εδώ είναι ότι η Ρωσία πιέζει για ξεχωριστή τριμερή συμφωνία η οποία θα υπογραφεί όταν τεθεί σε λειτουργία η Ουκρανική FTA. Και προέρχεται από το πεδίο εφαρμογής ε, της, ε, της FTA. Η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την πιθανή συμφωνία ως μοχλό για να ελέγξει το ουκρανικό εμπόριο. Γι' αυτό δεν στηρίζεται η δική μας θέση. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Τον ε, Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος. Η εντολή της Κομισιόν ε, όμως περιορίζεται αυστηρά σε αυτά που προβλέπονται στη Συμφωνία του Μίνσκ όπου αναφέρονται μόνο τα παράπονα της Ρωσίας ε, στο πλαίσιο της NDCFTA. Παρότι έχουν συνεχιστεί για αρκετό καιρό οι διαπραγματεύσεις, ε, η Ρωσία φαίνεται να μην μπορούσε να καθορίσει επακριβώς τα προβλήματα της μελλοντική συμφωνίας. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε στενά το θέμα και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο ο κύριος Μπορέλη για την Τουρκία. Ε, Εγώ για το Καζακστάν θέλω να μιλήσω, Πρόεδρε. Γιατί με την Τουρκία, για την Τουρκία μιλήσαμε ήδη. Αν συμφωνείτε. Α, Κεντρική Ασία, βέβαια. Αυτό ήταν. Ας πάμε όμως στις Ηνωμένε Πολιτείες. Στις 2 Ιουλίου έγινε η συνεδρία της ομάδας παρακολούθησης ε, για την προετοιμασία του τρίτου γύρου, συζητήσεις για τις υπηρεσίες και κάποια ίσονα θέματα. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις νομίζω. και θα υπάρξει ενημέρωση το Σεπτέμβριο. Μαγκρέμπ. Συνάντηση 8 Ιουλίου. Ανταλλαγή απόψεων. Στα πλαίσια της Euromed. Για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τινησία. Τώρα θα πάμε στην Κεντρική Ασία και στο Καζακστάν. Κύριε Μπορέλη. Ναι, ευχαριστώ. 25 Ιουνίου έγινε η, το Monitoring Group, ε, μίλησε για την Κεντρική Ασία με ειδική εστίαση στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, χώρες που για διάφορους λόγους ήταν ε, αντικείμενο προσοχής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα. Ε, μιλούσαμε για την πρώτη συνεδρίαση. Πρώτη φορά αυτή η Επιτροπή δημιουργεί ένα monitoring group που θα ασχοληθεί με την Κεντρική Ασία. Θεωρείται απαραίτητο και επίγον για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθήσει τη δυναμική στην Κεντρική Ασία και να αλληλεπιδράσει με τις χώρες αυτές. Οι δύο χώρες που παρακολουθούμε είναι μόνο κάποιες από αυτές που, που απασχολούν το Monitoring Group της Κεντρικής Ασίας. Τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουμε την παρακολούθηση για των υπολείπων κρατών. Σε ό,τι αφορά το Καζακστάν, που είναι η πιο μεγάλη χώρα της Κεντρικής Ασίας, η κατάσταση και οι εμπορικές σχέσεις είναι ενδιαφέρουσε πολλές χώρες ε, είναι είτε εισαγωγή είτε εξαγωγή ή επενδυτές στις χώρες αυτές. Οι διαδικασίες για τις, την υπογραφή των συμφωνιών εταιρική σχέση ε, είναι σε τελική φάση μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων. Θα ε, επι, επιτείνουμε, θα εντατικοποιήσουμε και τις εμπορικές μας σχέσεις και γενικά τις σχέσεις με τη με τη χώρα αυτή η επιστολή που έστειλε η ε, Επίτροπος Μάτσομ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, τονίζει ότι θα πρέπει προσωρινά να τεθεί σε εφαρμογή το, η συμφωνία για να μην χάσουμε την καλή στιγμή και να μην καθυστερήσουμε τη χώρα και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή, ε, ελπίζει μάλλον η το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το διαπραγματευτικό κείμενο. Η θέση της Επιτρόπου είναι πολύ λογική. Το Καζακστάν έχει μεγάλες οικονομικές φιλοδοξίες θέλει να μετασχηματιστεί, να διαφοροποιήσει την οικονομία του, να αυξήσει τις επενδύσεις σε τομείς, στη ε, γενοτομία, στην ε, επιστήμες, στην ε, έρευνα και στην ανάπτυξη, καθώς και στην παιδεία, να κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως τη δημόσια διοίκηση, το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την λογοδοσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητε συνεργασίας με το Καζακστάν και υπάρχουν ε, και εξάλλου πολλές ενεργειακές δυνατότητες στην Κεντρική Ασία, όπως αναφέρει και το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση του Ουσμπεκιστάν τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όχι είναι πιο μικρή χώρα και έχει μικρότερο δυναμικό, αλλά έχει και λιγότερες δυνατότητες συνεργασίας με εμά σε οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς το Ουσμπεκιστάν συχνά συζητήθηκε από εμά λόγω του λεπτού θέματος ε, της του Βάμβακος και πιστεύω ότι ο κύριος Αρένα ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό γιατί το παρακολούθησε εκ του σύνοικης. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη εκεί και ο πρέσβης Νόρο ε, προσεκλήθη στην ομάδα παρακολούθησης, μας παρουσίασε την κατάσταση και με βάση και τις εκτιμήσεις του ILO θα υπάρξει μια βελτίωση στη χώρα και των συνθηκών ζωής. Ε, θα υπάρξει προοδευτική μηχανοποίηση της ε, γεωργίας της χώρας θα, προ... ιδιωτικοποιηθεί η σοδιά του βάμβακος και ο πρωτογενής τομέας ε, θα διευρυνθεί και θα στραφεί και στα οποροκυπευτικά και θα σταματήσει, θα μειωθεί εν πάση η παιδική εργασία και η καταναγκαστική εργασία και στη σοδιά του Βάμβακος. Εμείς ως Επιτροπή ΙΝΤΑ παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις ε, στο Ουσμπεκιστάν σε συνεργασία με το ILO, με το Διεθνές δηλαδή Γραφείο Εργασίας και με άλλους φορείς. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Μπέγκε θα πάρει τον λόγο σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την Κούβα. Πράγματι, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο σχετικά και σα ευχαριστώ για την απόφαση των συντονιστών να δώσετε σε μένα το θέμα αυτό όσον αφορά την εποπτική ομάδα. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση για την Κούβα σήμερα με εκπροσώπους ε, της εξωτερικής, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής και ανέφεραν φυσικά ότι βλέπουν κάποια πρόοδο να επιτελείται σε σχέση με τα κεφάλαια του εμπορίου και του πολιτικού διαλόγου, επίσης ε, για το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και διαβάσαμε ότι ο πρόεδρος Κάστρο της Κούβας έχει την πρόθεση μέχρι το 2020 50% των νοικοκυριών να καλυφθούν με πρόσβαση στο διαδίκτυο, ίντερνετ. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς οι δυνατότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών θα χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατισμού των δημοκρατικών εξελίξεων και θετικών αυτών τάξεων, ε, τάσεων όπως και από πλευράς άλλων χωρών, άλλων υπήρων γιατί η διασύνδεση με το διαδίκτυο ωφελεί στο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο με δημοκρατικό τρόπο οι πολίτες. Φυσικά για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βενεζουέλα είναι η πιο σημαντική εμπορική εταίρη της Κούβας είναι δεδομένο και ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρώπη οι εισαγωγές από την Κούβα και ιδίως γεωργικών προϊόντων και οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, ε, μηχανικός εξοπλισμός ε, και προϊόντα της ευρωπαϊκής τεχνολογίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Κούβα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για αυτά και υπάρχει περιθώριο για συνεργασία και για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικά αναφέρθηκε ότι η Κούβα δεν, δεν υπέγραψε το, τη Συμφωνία Κοτονού, όμως από την άλλη πλευρά <clears throat> βρίσκεται εκτός προγράμματος από το 2014 διότι βάσει των στατιστικών στοιχείων ε, εξαιρούντο. Πρέπει να δούμε τώρα ποια συνέχεια θα δοθεί, ε, διότι είδαμε τα στατιστικά στοιχεία και πρέπει μελλοντικά να δοθεί μια ε, ξεχωριστή εξειδικευμένη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα γίνει σε σχέση με τα θέματα εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κούβας. Είχε συρρυκνωθεί πολύ σημαντικά το ποσοστό των εμπορικών αυτών συναλλαγών ε, ε, κατά τα πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να δούμε λοιπόν ποια στοιχεία βρίσκονται πίσω από αυτές τις εξελίξεις. Δεν αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στα διεθνή οικονομικά ε, μέσα η Κούβα. Όσον αφορά όμως το εμπόριο αναφέρεται ότι σε σχέση με τις συμφωνίες διευκόλυνσης, ε, μεταδιευκόλυνσης του εμπορίου, όπως και θέματα ε, κοινωνικής προστασίας θα μπορούσαν να προαχθούν. Καθώς επίσης αναμένεται ότι η υποεξέλιξη ε, νέες, νέα τάση για τις ε, επιπτώσεις ε, που θα μπορούσαν να υπάρχουν δημοσιονομικά. Κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον φυσικά, κάνοντας λόγο για τα στατιστικά στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, είχαμε ένα πρόβλημα γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία τα οποία παρέχονται από τις αρχές της Κούβας σε σχέση για παράδειγμα με την ταυτότητα των αλλοδαπών επενδυτών εδώ τίθενται θέματα εχεμήθειας και προστασίας των επενδύσεων αυτών και σε σχέση με το τι γίνεται για τις επενδύσεις όσον αφορά την, ε, τον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χρήση αυτών των στοιχείων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, προσθήκη ότι θα πρέπει αυτό να είναι το πιο σύγχρονο μέρος των ε, ε, περιοχών της ε, Λατινικής Αμερικής καθώς επίσης και για την δημιουργία μιας εναλλακτικής δυνατότητας όπως εξετάζεται στην διόρυγα του Παναμά και με την δυνατότητα ενός εκατομμυρίου εμπορευματοκιβωτίων που θα μπορούσαν να διέρχονται και πρέπει να δούμε εδώ τις δραστηριότητες της Κίνας και της Ρωσίας σε σχέση με την Κούβα καθώς επίσης και την ε, ε, διαδικασία για την ε, μεταφορά αυτή καθώς επίσης αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία εξετάσαμε. Προσβλέπουμε σε νέα στοιχεία τα οποία θα μας διατεθούν. Επόμενη συνάντηση το Σεπτέμβριο και υπό την ανακυκλούμενη προεδρία από πλευρά της, ενώ, της Κεντρικής Αμερικής που είναι στα χέρια του Σαλβαδόρ τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε και περνάμε στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης. 21, διορθώνω, 21 της ημερήσιας διάταξης. Διάφορα. Δεν υπάρχει τίποτα. Επόμενη συνάντηση της ε, Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής, 31 ε, Αυγούστου. Καλές διακοπές, να περάσετε καλά. Και θα σας ξαναδούμε, θα ξανασυναντηθούμε αναζωογονημένοι τέλη Αυγούστου. Ευχαριστώ για... I don't want to take much